Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκα. Το σχέδιο εμερήσιας διάταξης σας στάλει στις 17 Σεπτεμβρίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Νομίζω ότι είχατε αρκετό χρόνο, χρόνο για να το διαβάσετε, γιατί είχε δημοσιευθεί ηλεκτρονικά. Το πρώτο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πούμε είναι η συνεδρίαση που κάναμε στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα 5η, εγώ μαζί με τους συντονιστές και το Συμβούλιο. Ήταν μια συνεδρίαση αρκετά χρήσιμη και σημαντική, κατά την άποψή μου, γιατί όχι μόνο καταφέραμε να συνεδριάσουμε μαζί με το Συμβούλιο, αλλά και να συζητήσουμε επί εάν θα ήταν άτυπη συνεδρίαση ή επίσημη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Εμείς είπαμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συνεδριάζουμε πάντα επίσημα, ε, αλλιώς πηγαίνουμε στο καφενείο ή στην πιτσαρία. Επομένως ήταν μια επίσημη συνάντηση, ό,τι και να λέμε. Κάτι άλλο σημαντικό για αυτή τη συνάντηση είναι ότι καταγράφαψαμε αν και με ανορθόδοξα μέσα, ότι το Συμβούλιο απάντησε τελικά. Βέβαια θα πρέπει να μπούμε στην ουσία πώς απάντησε, με ποιους όρους απάντησε, στα αιτήματα και πιέσεις του Κοινοβουλίου. Ο τρόπος που απάντησε ήταν ασυνήθις. Γιατί η απάντηση δόθηκε ουσιαστικά με την ε, ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. αυτό είναι σημαντικό παρόλα αυτά. Το Συμβούλιο είπε κατ' επανάληψη, μέσω κυρίω ε, του Σουηδού ε, πρέσβη και του αναπληρωτή γενικού γραμματέα, ότι δεν είναι σε θέση να δεσμευθεί συγκεκριμένα στο πώς θα μας ενημερώνει επίσημα. Είπαν πολλές φορές ότι είναι διατεθειμένοι βέβαια να συζητήσουν με την Κομισιόν και να απαντήσουν σε διευκρινήσεις, αλλά στα πλαίσια τέτοιων συζητήσεων, όπως αυτή που κάναμε τελευταίως, όπως αυτή που σας είπα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν, μπορώ να θεωρήσω ένα βήμα προς τα εμπρός, σε σχέση με το διέξοδο που υπήρχε πριν. Βεβαίως, το Συμβούλιο ήρθε εδώ στο Κοινοβούλιο για να συνετήσει την Επιτροπή, την Επιτροπή μας. Αλλιώς, αν δεν είχε έρθει, θα, είχαμε... θα το είχαμε μεμφθεί με πολιτικό τρόπο το Συμβούλιο. Ε, γιατί δεν θα είχε απαντήσει. Κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να σας πω για τη συνεδρίαση αυτή είναι ότι μετά τη συνάντηση οι συντονιστές συνεδρίασαν και ήμουν και εγώ παρόν και αποφασίσαμε να αναβάλουμε τη συζήτηση και την ψηφοφορία που προβλεπόταν αυτή τη βδομάδα για την απαλλαγή του 2007, ούτω ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στον εισηγητή, στον οποίο τώρα θα δώσω το λόγο, να μελετήσει με κάθε προσοχή τις απαντήσεις που έδωσε το Συμβούλιο. Όχι μόνο ο εισηγητής, αλλά και όλοι μας νομίζω ότι πρέπει να μελετήσουμε τις απαντήσεις του Συμβουλίου. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο για να αποφασίσουμε. Τώρα, η νομική δυνατότητα της αναβολής επιβεβαιώθηκε κατά αυτή τη συνάντηση με τους συντονιστές και αναλύθηκε και από τη γραμματεία, το οποίο μας είπε ότι όντως είναι δυνατόν από νομικής άποψης να αναβάλουμε την απόφαση. Επομένως, στα πρακτικά που σας εστάλησαν θα βρείτε και ένα χρονοδιάγραμμα για τις συζητήσεις που θα κάνουμε γύρω από την απαλλαγή του 2007. Αν συμφωνείτε βέβαια. Τώρα. Τώρα θα δώσω τον, το λόγο στον κύριο Σόντεργαρτ που είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως μας είπε ο Πρόεδρος, υπήρξαν κάποιες ε, σημαντικές εξελίξεις από την τελευταία μας συνάντηση. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι είναι πολύ θετική η εξέλιξη αυτή, την οποία πετύχαμε μόνο και μόνο γιατί αυτή η Επιτροπή, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, πρόταξε αραγές μέτωπο. Και γιατί διεκδικήσαμε μια διαδικασία με περισσότερη διαφάνεια και περισσότερες ευκαιρίες, αν θέλετε, για ανταλλαγή απόψεων. Για να εξετάσουμε τους λογαριασμούς πριν δώσουμε το OK. Για τα νέα μέλη, θα ήθελα να τονίσω ότι στις 23 Απριλίου δεν δώσαμε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Αρνηθήκαμε για δύο λόγους. Για την έλλειψη απαντήσεων στις ερωτήσεις μας από πλευρά Συμβουλίου και δεύτερον γιατί το Συμβούλιο δεν θέλει να μας συναντήσει καν απευθεία. Αυτή ήταν η θέση του Συμβουλίου τότε. Η πρόταση του Συμβουλίου το Σεπτέμβριο είναι να κάνουμε μια άτυπη συνάντηση. Όμως τώρα είδαμε μια αλλαγή σε αυτή την ε, στάση. Εν μέρη, όπως είπε και ο πρόεδρος, μας δόθηκαν κάποιες απαντήσεις, παρότι πολύ έμεσα. Την περασμένη εβδομάδα, όπως ξέρετε, συνεδριάσαμε με τους, ε, όπως είπε και ο πρόεδρος, με τους συντονιστές και με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, η έκθεση που ετοιμάστηκε για σήμερα δεν είναι επικαιροποιημένη. Εξαιτία του τρόπου που εργαζόμαστε στο, συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και λόγω των προθεσμιών της μετάφρασης, η μετάφραση γράφτηκε λίγες μέρες μετά την εκλογή, μετά τις Επομένως, χρειαζόμαστε μια νέα έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις που είχαμε τελευταίως. Και μια έκθεση που θα λέει ότι το θέμα αυτό θα αναβληθεί από την Ολομέλεια του Οκτωβρίου θα πάει στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Πρέπει να γράψουμε μια επίσημη επιστολή στο... Ε, από πλευρά ε, Κοινοβουλίου και θα πρέπει να την εγκρίνει και ο Πρόεδρο. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε αυτέ τι συζητήσει στο συντομότερο δυνατόν. Αύριο, ίσω. Γι' αυτό λοιπόν θα έχω ένα νέο σχέδιο για μια νέα έκθεση, το οποίο θα στείλω στους κοιόδες εισηγητές ούτως ώστε να ακούσουμε σχόλια. Επίσης είμαι έτοιμος να συναντήσω και τους κοιόδης εισηγητές. Ούτως ώστε να διατηρήσουμε αυτή τη σχεδόν ομόφωνη στάση που είχαμε από την αρχή της διαδικασίας, χάρη και στην οποία πετύχαμε τα θετικά αποτελέσματα που πετύχαμε. Επομένως, ποια, είναι, ποια θα είναι η θεμελιώδης αρχή στην έκθεσή μου η κατευθυντήρια αρχή. Από τη μία, θα καλωσορίζουμε το γεγονό και θα εκφράσουμε την ικανοποίησή μα ότι το Συμβούλιο επιτέλου απάντησε στι ερωτήσει μα και συναντήθηκε με του εκπροσώπους τη Επιτροπή μα. Αυτή η θετική εξέλιξη όμως θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Από την άλλη, θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό που λέγαμε στην εκθεσή μας. Πάντα λέγαμε κάτι τέτοιο, ότι για να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να εγκρίνουμε τους λογαριασμούς, αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον το Συμβούλιο θα πρέπει ετησίως να υποβάλει έκθεση δραστηριοτήτων, κάτι που όλα τα υπόλοιπα ε, θεσμικά όργανα στέλνουν στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή το Συμβούλιο στο μέλλον θα πρέπει να απαντάει στα γραπτά ερωτήματα που υποβάλλουμε και να απαντάει στον πρόεδρο της Επιτροπής μας. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο στο μέλλον θα πρέπει να είναι σε θέση και σε ε, διάθεση να μας συναντήσει για να συζητήσουμε τους λογαριασμούς του. Αυτό έχει να κάνει όχι με επίσημα στοιχεία, με επίσημα και τυπικά χαρακτηριστικά, για να μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή θα πρέπει να λέμε τι περιμένουμε από το Συμβούλιο. Λοιπόν, αύριο θα έλεγα να εγκρίνουμε λοιπόν τους λογαριασμούς, αλλά να παραμείνουμε μετακίνητοι για την έγκριση και την απαλλαγή του 2008. Τώρα, για τις απαντήσεις που λάβαμε από το Συμβούλιο, υπάρχουν μεταξύ αυτών κάποιες καλές απαντήσεις, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες είναι αβάσιμες, ασταθείς. Και κάποιες απαντήσεις που πρέπει να επεξηγηθούν περαιτέρω. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στη διαδικασία που έχουμε τώρα αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δώσουμε απαλλαγή. Θα πρέπει να σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την έκθεση για να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχουν ασαφείς περιοχές που θα θέλαμε να τις είχαμε εξετάσει περαιτέρω και θα ζητάμε ε, από τον εισηγητή του 2008 να διερευνήσει περισσότερο αυτά τα στοιχεία ακριβώς, αυτά τα σημεία, αυτές τις περιοχές. Το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι κάτι για την κατάσταση που βασιλεύει στο Συμβούλιο. Φυσικά υπάρχουν διεστάμενες απόψεις για την κατάσταση στο Συμβούλιο. Αλλά από τις πληροφορίες που εγώ τουλάχιστον έχω, ορισμένοι ήταν εναντίον της δημοσίευσης των απαντήσεων σε μας ε, στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Όμως τελικά δεν χρειάστηκε να δοθεί σκληρή μάχη στο Συμβούλιο για να δημοσιευθούν αυτές οι απαντήσεις. Υπήρχε τελικά μια ευρεία υποστήριξη υπέρ του να γίνει από πλευρά του Συμβουλίου και ένα βήμα παραπάνω για να εξασφαλιστεί ένα άνοιγμα και η διαφάνεια από πλευρά Συμβουλίου. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Συμβούλιο γι' αυτό λοιπόν. Αλλά χάρη σε αυτό μπορεί να γίνει και η δική μας δουλειά, χάρη σε αυτή τη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Φυσικά δεν είναι εδώ ο χώρο να υψέλθουμε στα επί της ουσίας. Ο εισηγητή απλά μια αναφορά έκανε. Αν συμφωνείτε λοιπόν η συζήτηση για την ψηφοφορία αναβάλλεται για την συνεδρίαση της 3 η και 4 η Οκτωβρίου για να ψηφιστεί κατόπιν στην Ολομέλεια στις 26 και 27 Νοεμβρίου. Αν συμφωνείτε αυτή τη διαδικασία είχαμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε και στην συνεδρίαση των συντονιστών. Στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε την έγκριση των πρακτικών, τα οποία σας απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 22 Σεπτεμβρίου του 2009. Ο γραμματέας εδώ μου επισημαίνει ότι για σήμερα το απόγευμα υπάρχει ένα πρόβλημα για την μετάφραση στα βουλγαρικά, η οποία δεν είναι έτοιμη. Έχει προβλεφθεί όμως για αύριο. Έχετε και μία σειρά από ανακοινώσεις, ε, δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο, νομίζω ότι τα διαβάσατε, έχουμε το web streaming, το εγχειρίδιο του 2009... Κάτι σημαντικό είναι η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Και για αυτό το σημείο θα πρέπει να σας ε, αναφέρω περιληπτικά μια πολύ δύσκολη εντό εισαγωγικών διαπραγμάτευση η οποία έγινε τις τελευταίες ημέρες με το ελεγκτικό συνέδριο για να προσπαθούμε να εξεύρουμε μια λύση η οποία θα μπορέσει να καλύψει και κάποιες απαιτήσει οι οποίες ε, για να είναι, πω την αλήθεια είναι και λίγο ε, υπερ, υπερβολικές, δηλαδή ήταν περισσότερες οι απαιτήσει ε, για αυτόν που εκτυπώνει την έκθεση και όχι για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα μακρηγορήσω, έγιναν συναντήσεις ε, αρκετά κουραστικές. η λύση στην οποία καταλήξαμε, η οποία λίγο πολύ καλύπτει και όλες τις ανάγκες, είναι ότι η συζήτηση για την έκθεση θα γίνει την 3η 10 Νοεμβρίου 2009. Θα βρείτε και ένα χρονοδιάγραμμα με ωράρια, το οποίο έχει καθορίσει η γραμματεία και λαμβάνει υπόψη διπλές ανάγκες. Τη δική μας την απέτηση, η οποία κατά την άποψή μου είναι προτεραιότητα, που είναι να κάνουμε μια εις συζήτηση της έκθεσης και να μπορέσουμε να θέσουμε και ερωτήσεις ε, ή να ζητήσουμε και κάποιες διευκρινήσεις ε, στους, στα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου και κατόπιν υπήρχε και μία απέτηση που κατά την άποψή μου είναι δευτερεύουσα αλλά φαίνεται ότι για το ελεκτικό συνέδριο είναι απέτηση προτεραιότητας. Αυτοί μέχρι το 12 το μεσημέρι θέλουν να δημοσιοποιήσουν στον τύπο το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Μία ακόμα πτυχή είναι το γεγονός ότι η έκθεση θα είναι διαθέσιμη και θα διανεμηθεί την προηγούμενη, στις 9 Νοεμβρίου γύρω στο μεσημέρι. Και στις 6 του μηνός που είναι Παρασκευή, θα δοθεί ένα αντίγραφο στον πρόεδρο και στον εισηγητή. Μέχρι τη Δευτέρα πάντως σίγουρα θα την έχετε στη διάθεσή σας όλοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί την επόμενη μέρα, την Τρίτη, ε, θα μπορούμε να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και να έχουμε και μια σαφή εικόνα της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Ένα ακόμα σημείο στο οποίο υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ ημών και του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν το κατά πόσον η συνεδρία θα γίνει και κλεισμένων των θυρών ή θα είναι ανοιχτή σε όλους. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτή η συνεδρία θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους για λόγους διαφάνειας, διότι δεν υπάρχει και τίποτα το οποίο να είναι εμπιστευτικό και σε αυτό λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα, διότι στην τελευταία επιστολή που μου διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επ' αυτού, επομένως ε, Ελπίζουμε να μην ε, υπαναχωρήσουν στο σημείο αυτό. Στη συνέχεια θα δείτε ότι έχουμε τις ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε, και την ετήσια διάσκεψη του IAS. Ένα ακόμα σημείο το οποίο θα ήθελα να σας επισημάνω, ε, το οποίο μπορεί και να μην μας ε, είναι απαραίτητο, είναι να θυμηθείτε να φέρετε τις κάρτες σας αύριο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Στο σημείο 4 τώρα έχουμε τις συστάσεις των συντονιστών της τελευταίας συνεδρίασης που κάναμε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2009. Δεν θα τα διατρέξω αυτά, διότι έχετε λάβει όλοι το σχετικό σημείωμα, αλλά υπάρχει ένα προκαταρκτικό ζήτημα πολύ σημαντικό, το οποίο το συζητήσαμε και στην αρχή της συνεδρίασης της 10 Σεπτεμβρίου με τους συντονιστές, που είναι το θέμα της συμμετοχής των μη εγγεγραμμένων ευρωβουλευτών στη συνεδριάση των συντονιστών. Εδώ θα πρέπει να σας ενημερώσω και για το τι αποφάσισε η διάσκεψη των προέδρων στην οποία συμμετείχα. Δεν υπάρχουν ακόμα τα πρακτικά, αλλά να σας πω εκ των προτέρων ότι η ομόφωνη απόφαση των προέδρων όλων των επιτροπών είναι οι μη εγγεγραμμένοι ευρωβουλευτές να μην μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδριάση των συντονιστών. Εκτός και για την περίπτωση στην οποία θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιο τρόπο που θα διαφυλάσσουν το δικαίωμα των Ευρωβουλευτών να ε, μπορούν να πληρώσουν ε, τις υποχρεώσεις τους. Επομένως, ε, έμεινε η εκκρεμότητα να θέσουμε και το θέμα στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Νομίζω ότι στη συνεδρίαση των συντονιστών η πλειοψηφία των συμμετοχόντων ήταν αντίθετη. Μιλάω για τις συνεδρίες των συντονιστών ε, της δικής μας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Οι περισσότεροι λοιπόν είπαν ότι ήταν αντίθετοι. Διαβάσαμε και την ε, συνθήκη η οποία κατά γράμμα λέει ότι δεν υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής ε, στη συνεδριά των συντονιστών για τους μη εγγεγραμμένους ευρωβουλευτές. Επειδή όμως ε, δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση και επειδή το θέμα είναι και σχετικά ευαίσθητο, αποφασίσαμε να σας υποβάλουμε το ζήτημα και στην ε, σημερινή συνεδρίαση, να ψηφίσουμε και να εκφραστεί άποψη της Επιτροπής μας. Το συζήτησα και με τη γραμματεία και επιτρέψτε μου να σας προτείνω μία λύση η οποία λαμβάνει υπόψη της και αυτή την απόφαση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Οι ευρωβουλευτέ που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε πολιτικέ ομάδε δεν μπορούν να συμμετέχουν σε συνεδριάσει των συντονιστών. Θα πρέπει ίσω να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση που θα του επιτρέπει να ενημερώνονται κατά κάποιο τρόπο για το τι συμβαίνει. Μια λύση θα ήταν στα μέλη ή στο μέλος, ε, διότι μπορεί να συμμετέχει ένας ε, που δεν είναι και γραμμένα σε πολιτικές ομάδες, να λαμβάνουν το σημείωμα των συντονιστών, την ημερήσια διάταξη αν θέλετε της συνεδρίασης που θα κάνουν οι συντονιστές, γιατί έτσι θα τους επιτρέπεται να είναι ερημερωμένοι και ταυτόχρονα να μπορούν ε, ίσως μέσω των συντονιστών ή μέσω του Προέδρου να προσθέτουν την άποψή τους. Όσον αφορά το αποτέλεσμα της συνεδρίασης των συντονιστών, το κάθε μέλος θα έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για το τι αποφασίστηκε, όπως συμβαίνει και με όλα τα υπόλοιπα μέλη των, ε, της Επιτροπής. Εάν ε, ε, συμφωνείτε με αυτό, εκτός και αν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, σήμερα θα πρέπει να αποφασίσουμε, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να μπορούμε να έχουμε και μια σαφή εικόνα για το τι θα κάνουμε. Παρακαλώ. Πρόεδρε, είμαι αντίθετος με αυτή την πρόταση γιατί υπάρχει ένας κανόνας στο Κοινοβούλιο για τους συντονιστές και δεν θέλω από την πλαϊνή πόρτα, από ένα παρασυράκι, οι συντονιστές να ακούγονται περισσότερο μέσω της γραμματείας της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού από ότι εμείς. Ε, έτσι καλώς εκπροσωπούνται μέσω της γραμματείας. Μία πολιτική ομάδα είναι μία ομάδα και οι συντονιστές δεν αποτελούν πολιτική ομάδα. Εγώ δεν συμφωνώ διόλου με αυτή την πρόταση. Η μία εγγεγραμμένη, η μία εγγεγραμμένη, συγγνώμη, μπορείτε να τους πείτε ό,τι θέλετε, ε, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία που προτείνεται για τους μία εγγεγραμμένους ε, συμφωνεί με το καταστατικό και τους κανόνες λειτουργία του Κοινοβουλίου, διότι θα μπορούν να εισέλθουν μέσα από ένα παραθυράκι και μέσω της γραμματείας. Πιστεύω ότι η γραμματεία ε, της Επιτροπής Ελέγχου δουλεύει για όλου μα και αν δεν υπάρχει υπάρχει κανένας μη εγγεγραμμένος στους συντονιστές, ε, τι να κάνουμε, ας μην υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να πούμε πλαγίως ε, μέσω συντονιστών. Μπορούμε, μπορούμε να τους δώσουμε την ατζέντα, την ημερήσια διάταξη, εντάξει, να ενημερώνονται για την ημερήσια διάταξη και τα θέματα, αλλά όχι να μπουν από ένα παραθυράκι. Όχι πλαγίως ε, με τον τίτλο του συντονιστή. Και, και εγώ ε, ομολογώ ότι ως εκπρόσωπος της χώρας μου, ε, εντάξει, ας μην πα, πα, παρετούμε από αυτό το δικαίωμα. Μα το ίδιο λέμε. Νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε ότι μπορούν να έχουν την ημερήσια διάταξη. Έτσι δεν είναι. Ναι. Την ημερήσια διάταξη. Συνένει η κυρία. Βεβαίω, ωραία. Τότε συμφωνούμε. Ναι, μία άλλη ερώτηση ακόμα, για να μην ε, υπάρχει σύγχυση εσείς πρόεδρε είπατε τα εξής από ό,τι κατάλαβα ότι οι μη τα μη εγγεγραμμένα μέλη όχι μόνο θα λαμβάνουν την ημερήσια διάταξη αλλά και θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω της γραμματείας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά διότι αφενός θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα η μία εγγεγραμμένοι που είναι μέλη της Επιτροπής να ενημερώνονται για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ε, στη συνεδρίαση των συντονιστών. Όμως, η έκφραση γνώμης, η γνωμοδότηση δηλαδή, αλλάζει τα πράγματα, διότι τότε θεωρητικά μπορεί να προκύψει το εξής. Ένας μία εγγεγραμμένος να εκφράσει τη γνώμη του μέσω της γραμματείας επί της συνεδριάσεως. Δηλαδή, θα εκφράσει τη γνώμη του για ένα θέμα στην ε, ημερήσια διάταξη. Οπότε κυρία Γκρέσλε θα έχει δίκιο. Ε, ε, θα εισέρχονται πλαγίως, θα δημιουργηθεί ένα παραθυράκι. Το να μην ενημερώνεται για την ατζέντα, εντάξει, δεν είναι σωστό να τους δώσουμε την ατζέντα και να ξέρουν για να μπορούν να προετοιμαστούν για τις εργασίες της ομάδας μας. Εκεί δεν έχω, της επιτροπή μας, συγγνώμη. Κοιτάξτε, συζητήσαμε ακόμη και στη διάσκεψη των Προέδρων να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε αυτές τις απαιτήσει. Δηλαδή, όχι να τους επιτρέψουμε να συμμετάσχουν, αλλά να τους δώσουμε έναν τρόπο για να τους κάνουμε με κάποιο τρόπο ε, ενήμερους μέτοχους. Δηλαδή, να δίνουμε την ημερήσια διάταξη, όχι για να εκφράζουν γνώμες ή αξιολογήσεις επί της συνεδρίασης. Με την ημερήσια διάταξη μπορούν να ασκήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματά τους. Αλλά στη συνεδρίαση των συντονιστών προφανώς δεν, συνε... δεν συμμετέχουν. Ούτε άμεσα ούτε έμεσα μέσω άλλων. Μέσω της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γράψουν, ας πούμε, αν θέλουν, μετά μια επιστολή, έτσι. Αυτό εννοούσα. Δεν θέλω να τους δώσω το δικαίωμα εμέσως να συμμετέχουν στη συνεδρία των συντονιστών, έτσι. Ε, Επομένως, συμφωνούμε. Στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών θα συμμετάσχουν μόνο οι συντονιστές που προέρχονται από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Εν αναμονή των πρακτικών της συνεδρίασης της 15ης ε, Σεπτεμβρίου της διάσκεψης των Προέδρων και ε, κάποιων ε, γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων που θα μπορούσαν να εμφανίσουν άλλα σενάρια ενημέρωσης ή συμμετοχής των μη εγγεγραμμένων, μένουμε σε αυτά που είπαμε. Τώρα, για το σημείο 5, αυτό όπως σας είπα δεν θα το συζητήσουμε σήμερα, το αναβάλουμε. Για τις 23 Οκτωβρίου. Και τώρα. Πάμε στο σημείο 6. Έχουμε την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, της Όλαφ. Για την για τη δραστηριότητα, την οικονομική δραστηριότητα 31 Δεκεμβρίου 2000 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008. Ο κύριος Φρανς Μπρούνερ, Γενικός Διευθυντής της ΟΛΑΦ, θα μας παρουσιάσει αυτή την ε, έκθεση και εν συνεχεία μετά την παρουσίαση ή οσδήποτε θέλει διευκρινήσεις ή θέλει να θέσει ερωτήσεις μπορεί να το κάνει. Prego, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ καταρχάς θερμά που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την έκθεση δραστηριοτήτων της Όλαφ του 2008. Πριν σας παρουσιάσω την έκθεσή μου, μου επιτρέπετε μερικές γενικές παρατηρήσεις ιδιαίτερα επειδή η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού έχει νέα μέλη, τα οποία δεν ήταν παρόντα πέρσι και ε, το θέμα μας αυτό είναι οπωσδήποτε περίπλοκο και πολύ πυκνό, πολύ πυκνή αυτή η έκθεση δραστηριοτήτων. Είναι λοιπόν ε, ε, δυσκολοχώνευτα θέματα αυτά, γιατί αφορούν περιπτώσεις ε, των οποίων δεν ξέρουμε το υπόβαθρο και το ιστορικό. Η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού είναι ένα σημαντικό εταίρος και συνεργάτης για την Όλαφ, για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς και της απάτης μέσα στα πλαίσια ελέγχου του προϋπολογισμού. Η συνεργασία με το εξήκο κοκομπού και ΟΛΑΦ έχει βελτιωθεί εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως άρχισε η συνεργασία αυτή κάπως θυελωδός, αλλά αναπτύχθηκε ομαλά και πολύ ε, επικοδομητικά τα τελευταία χρόνια και προς όφελος της προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ατασταλίες και απάτες. Είμαι απολύτως πρόθυμος και εγώ έχω εκφράσει επανειλημμένα στην προσωπική μου βούληση για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας. Βλέπω εδώ ορισμένα νέα πρόσωπα αλλά και πολλά νέα μέλη και γι' αυτό θα κάνω ακόμα μερικές παρατηρήσεις. Από την αρχή του 2000 ε, είμαι διευθυντής ε, του Όλαφ ε, και έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη του οργανισμού. Δέκα χρόνια γιορτάζουμε λοιπόν φέτος και η Όλαφ έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν αξιοσέβαστο και αναγνωρισμένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Είμαι λοιπόν υπερήφανος ε, διότι καταφέραμε αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα και δεν έχουμε καθόλου παρατηθεί από τις προσπάθειές μας. Το Όλαφ υπόκειται βεβαίως σε ορισμένους περιορισμούς μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Μπορεί να εκτελεί διοικητικούς ελέγχους και έρευνες, αλλά δεν είναι υποχρεωτικές. Η ετήσια έκθεση του βεβαίως υπόκειται στον έλεγχο του δικαστηρίου, αλλά εκδίδει το όλαυ συστάσεις στις εθνικές αρχές και του εθνικούς φορείς ή στις γενικές διευθύνσεις για τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόσουν και τι επιπτώσει τους. Και βεβαίω, το η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ποιοτική μας εργασία, η προβολή της ποιότητα. Θα ήθελα λοιπόν Καταρχά να διαβεβαιώσω όλους σας και τον πρόεδρο κύριο Ντεμαγκίστοης ότι θα ήταν μια μπασαυμάση ευκαιρία τα νέα μέλη του Κοκομπού να επισκεφθούν τα γραφεία της Όλαφ την έδρα μας για να διαμορφώσουν μόνοι τους μια εικόνα συνολική των δραστηριοτήτων μας. Ε, η Τόλαφ ε, είναι ένα περίπλοκο όργανο και έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουν τα νέα μέλη όλες τις περίπλοκες πτυχές της εργασίας μας και της ευθύνης μας. Τώρα, όσον αφορά το, την έκθεση δραστηριοτήτων μας και τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, δείχνουν ότι το Όλαφ λειτουργεί απολύτως αντικειμενικά και ανεξάρτητα. Θα σας πω μερικές, ε, μερικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην έκθεση του 2008. Οι, οι φάκελοι τους οποίους ε, εξετάσαμε ε, αυξήθηκαν από χρόνο σε χρόνο και τα τελευταία χρόνια είχαμε 55% αύξηση των ε, ύποπτων περιπτώσεων προς εξέταση και περισσότερες από χίλιες Είχαμε ε, από χίλια, ε, πήρε πάνω από χίλια σήματα να ερευνήσουμε μια ΑΒ υπόθεση. Μας ε, ειδοποίησαν δηλαδή ότι κάπου κάτι συμβαίνει. Τα τελευταία πέντε χρόνια ε, ο αριθμός των ε, περιπτώσεων που άνοιξαν, οι φάκελοι που ανοίχτηκαν, ε, αυξήθηκαν σημαντικά και το 2008 ήταν 204 φάκελοι. Βεβαίως δεν είναι μόνο ο αριθμός των φακέλων και των υποθέσεων, αλλά και τα αποτελέσματα. Ιδιαίτερα πώς παίρνουμε πίσω τα λεφτά τα οποία παρανόμως έχουν δαπανηθεί. Εξετάζουμε λοιπόν και το δημοσιονομικό follow-up, δηλαδή τη συνέχιση των υποθέσεων και 450 ε, εκατομμύρια ευρώ συλλέχθηκαν το 2008, ουσιαστικά δηλαδή επιστράφησαν εκεί όπου, από όπου δεν θα έπρεπε να είχαν βγει ή ήταν το αποτέλεσμα της ε, της έρευνάς μας για τις απάτες και τις ατασταλίες και το, το ότι σπράξαμε, καταφέραμε να, να επιστρεφεί ένα τέτοιο τεράστιο ποσό παρά τον προϋπολογισμό των 50 εκατομμυρίων ευρώ δείχνει ότι αξίζουμε τα λεφτά μας. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στον ποινικό τομέα μου. Εδώ καταδικάστηκαν 300 άνθρωποι από τα εθνικά δικαστήρια, ε, τα ποινικά δικαστήρια δηλαδή, που είναι ένας αρκετά μικρό αριθμός σε σχέση με τα 10 χρόνια δραστηριοτήτων μας. Όμως αυτό δυστυχώς ε, οφείλεται στο ότι δεν είναι και άριστη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών και ελπίζω οι περισσότερες υποθέσεις που άνοιξαν μετά τη δική μου προεδρία να μπορέσουν και να κλείσουν το ταχύτερο διότι 10 χρόνια είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα για να καταφέρουμε να καταδικαστεί κάποιος ποινικά. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την κυρία Γκρέσλε για αυτό το σεμινάριο συνεργασίας που οργάνωσε ε, με το Κοκομπού το Φεβρουάριο του 2009 πρέπει να συνεχίσουμε και να επιδιώξουμε την καταδίκη όλων αυτών που έχουν παρανομήσει και των καταχραστών. Και αυτό το σεμινάριο Κοκομπού ήταν πάρα πολύ επιτυχές. Η... Τα αποτελέσματα και επιτυχίες του Όλαφ δεν μπορούν να παρουσιαστούν μόνο με στατιστικά στοιχεία, αλλά πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και στην πρόληψη των απατών. Στο πλαίσιο αυτό το 2006 ξεκινήσαμε διάφορα προγράμματα πληροφόρησης όπως το πρόγραμμα Πλούτο, ε, πληροφορίας λογιστικής φύσεως της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, Πληροφοριών Ινφσο, επίσης το πρόγραμμα Διαφανή Ενίσχυση Trade, ε, στο θέμα της εξωτερικής βοήθειας, δηλαδή διαφάνεια ε, στα κονδύλια τα οποία δίδονται εξωτερική βοήθεια και ανάλυση ρίσκου για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης. Πού εστιάζουμε τώρα τις δραστηριότητε μας. Καταρχάς, οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν ένα μικρό αριθμό κρατών το 2008 ασχοληθήκαμε με έξι κράτη-μέλη. Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, Βρετανία. Ε, αυτές οι χώρες κάλυψαν το 55% των περιπτώσεων από συνολικά 204. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως αναγκαίο ότι αυτές οι χώρες συγκεκριμένα έχουν περισσότερες απάτες, εκεί συμβαίνουν περισσότερες απάτες. Αντίθετα σημαίνει ότι εκεί έχουμε μια καλύτερη συνεργασία και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Οπότε μπορούμε και εντοπίζουμε και επιλύουμε ε, περιπτώσεις απάτης. Ε, έχουμε και άλλε χώρε όπου σημειώνονται απάτες και παρανομίες, αλλά δεν ε, δηλώνουν ή δεν συντάσσουν εκθέσεις ε, για τις απάτες αυτές. Δεν ε, θέλω να πω ούτε να κατηγορήσω συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Παντού προσέχουμε και έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Επίσης, έχουμε εντατικοποιήσει τη συνεργασία μας με τις βουλγαρικές και ρουμανικές αρχές, τους αρμόδιους φορείς για την καταπολέμηση της απάτης και είναι πάρα πολύ ψηλά στην εμμυρίση διάταξή μας αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία. Έχουμε μάλιστα και την ομάδα δράσης Βουλγαρίας. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας είναι να βοηθήσουμε τα κράτη αυτά να αυτοβοηθηθούν, δηλαδή να μπορούν να λύσουν από, μόνο, από μόνες τους οι χώρες αυτές τα προβλήματα με τους δικούς τους συνεργάτες, να μπορέσουν δηλαδή να τσεκάρουν την κατάσταση μέσα στα εθνικά του σύνορα. Έχουμε επίσης, ε, διάφορες, έχουμε επίσης συνεργαστεί επανειλημμένως με πολλές ε, τελωνιακές αρχές, τις οποίες υποστηρίξαμε, βοηθήσαμε το 2008 και έχουμε επίσης συνυπογράψει μία, ένα συμφωνητικό, μία σύμβαση συνεργασίας με μία μεγάλη εταιρεία παρασκευής τσιγάρων, δεδομένου ότι εκεί ακριβώς παρουσιάστηκε ένα μεγάλο πρόβλημα απάτης. Θα συνεχίσουμε να βοηθούμε την ε, καπνοβιομηχανία, στην καταπολέμηση της ε, απάτης και ε, προσπαθούμε να βρούμε καλύτερα μέτρα καταπολέμησης και πιστεύω ότι η εργασία την οποία κάνουμε είναι πάρα πολύ καλή διότι ναι μεν πολλοί φάκελοι οδηγούν στην ποινική δίωξη αλλά το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στις ε, ε, διοικητικές ε, διαδικασίες τις οποίες παρακολουθούμε και ενισχύουμε τους εταίρους μας. Προσπαθούμε λοιπόν να ενισχύσουμε τις διοικητικές τους υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν τις απάτες και να τις διώξουν ποινικά. Συνεργαζόμαστε βεβαίως και με την Europol και με την Eurojust. Έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μας αλλά και με διεθνείς οργανισμούς, με διεθνείς ε, φορείς όπως ε, τα Ηνωμένα Έθνη και με τρίτες χώρες. Έχουμε εντατικοποιήσει λοιπόν τις συνεργασίες μας με όλους τους ε, συναρμόδιους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα διεθνώς. Και πιστεύουμε ότι πολλοί, φορείς, ε, ε, ε, έχουν, έχουμε ενισχύσει, έχουμε βοηθήσει πολλούς φορείς με αποτρεπτική δράση, οι οποίοι έχουν ενεργήσει παραδειγματικά και έτσι έχουν επίσης πολλούς απατεώνες ότι μην αγγίζετε αυτό τον τομέα, μην προσπαθήσετε να κάνετε κάποιο λαθρεμπόριο, γιατί έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και προσέχουμε συνεχώς τι κάνουμε. Επίσης, το θέμα της εξωτερική βοήθειας, το οποίο είχαμε συζητήσει και πέρσι, πρέπει να συγκεντρωθούμε περισσότερο στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις και καλύπτουμε όλο και περισσότερες, όλο και μεγαλύτερες περιοχές ε, του κόσμου και ιδίως σε ε, σοβαρές περιπτώσεις το 70% των πόρων μας καλύπτει ακριβώς αυτές τις πολύ σοβαρές περιπτώσεις και σε άλλες υπήρους και παρακολουθούμε ε, από το 2008 όλα αυτά τα πειθαρχικά και τα πειθαρχικά μέτρα τα οποία έχει επιβάλει η Κομισιόν βάσει των φακέλων τους οποίους έχουμε ξεκινήσει εμείς. Έχουμε εφαρμόσει την αρχή της μηδενικής ανοχής ε, έναντι των απατών και των ατασταλιών σε όλα τα όργανα επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά τις περιπτώσεις ε, διαφθοράς και απάτης και τη σωστή εφαρμογή των μηχανισμών δίωξης. Παρόλο που οι περιπτώσεις μας είναι πολύ περίπλοκες, το 2008 καταφέραμε να μειώσουμε τον χρόνο χειρισμού ενός φακέλου το 2008 ήταν ε, η δραστήρια φάση, η ενεργός φάση χειρισμού φακέλου, ε, μειώθηκε από 28 σε 24 μήνες. Καταφέραμε λοιπόν μία σύντμηση, μία σμίκρυνση της περίοδου χειρισμού ενός φακέλου και αυτό το καταφέρουμε στο 60% έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το βουνό των φακέλων που έχουμε πάνω στα γραφεία μας. Και τέλος, όσον αφορά την πολιτική των ανθρώπινων πόρων, εμείς έχουμε περίπου 475, συνολικά 475 συνεργάτες και εδώ έχουμε σταθεροποιήσει τον αριθμό των συνεργατών μας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν 475 και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο ξανά που με τον διορθωτικό προϋπολογισμό 2008 κατάφερε να τον εγκρίνει ταχύτατα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και εμείς τις διατάξεις ε, στο προσωπικό μας και να επιβάλλουμε μια σταθερότητα ε, και μια ποιοτική εξασφάλιση και εμπειρία ε, στην επιλογή του προσωπικού μας και στις προσλήψεις σε άλλες ε, υπηρεσίες ε, το προσωπικό συνέχεια αυξάνεται. Σε εμά ε, πιστεύω ότι οι, ποιοτικέ μας, οι ποιοτικές μας επιλογές, παρόλο η κατάσταση στην αγορά από απόψεως ποιότητος είναι δύσκολη, ήταν πάρα πολύ καλή και προσβλέπουμε προσβλέπουμε και στο μέλλον στην υποστήριξη μέτρων που θα αναπτύξουν περισσότερο το προσωπικό μας, δηλαδή μετεκπαίδευση, επιστημονική εκπαίδευση κλπ. Γενικά πρέπει να πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή στελέχωση για να μπορέσουμε να έχουμε τα ίδια θετικά αποτελέσματα και την επόμενη δεκαετία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, ο κ. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα Σας καλωσορίζω στην Κοκομπή. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες εξηγήσεις ε, για την κατάσταση στη Βουλγαρία. Στην προηγούμενη ε, κοινοβουλευτική θητεία, αυτή εδώ η Επιτροπή ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το θέμα και ειδικά σε ό,τι αφορά την απαλλαγή. Και με ορισμένου ε, συναδέλφους και μαζί σας είχαμε χωριστές συνεδριάσεις στις αρχές του χρόνου. Ήδη στις αρχές του χρόνου μας δώσατε την ε, εντύπωση ότι οι βουλγαρικές αρχές ασχολούνται πολύ αυστηρά με το θέμα. Παραδείγματο χάρη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ασχολείται ειδικά με την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Εσείς μας είχατε πει ότι είχατε την εντύπωση πως τα πράγματα εξελίσσονταν θετικά στη Βουλγαρία. Εν συνεχεία έγιναν ε, εκλογές στη Βουλγαρία, προέκυψε μια νέα κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί τα ποσά είναι ψηλά. Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά το δικό μα θεσμικό όργανο. Πριν από λίγες εβδομάδε κυκλοφόρησαν κάποιες εκθέσεις για το γεγονός ότι ο Μεσουλαδητή είχε πάρει μία απόφαση σε ό,τι αφορά το θέμα ενό δημοσιογράφου, ο οποίο ήθελε να έχει πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούσαν πιθανές ε, παρατυπίες, ειδικά για την ε, οικοδόμηση αυτού του κτηρίου, στο οποίο βρισκόμαστε, και του διπλανού κτηρίου. Ε, και τότε μιλήσαμε και για την κατάσταση, την στάση, αν θέλετε, και την συμπεριφορά της Όλαφ. Κύριε Μπρούινερ, θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα λόγια για το ρόλο της Όλαφ. Τι πιστεύετε εσείς για αυτή την υπόθεση, για την απόφαση του διαμεσολαμητή. Κύριε Μπρούινερ, παρακαλώ. Äh, äh, Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, Έχουμε μια επαρκή στελέχωση. Είναι πολλοί συνεργάτες μας, αλλά χρειάζονται για να προχωρήσουμε. Η παλαιά διοίκηση, ιδιαίτερα στο διοικητικό τομέα, μπόρεσε να περάσει πολλές ε, αλλαγές και πιστεύω ότι Ιδίω τώρα που ε, έχουμε την ε, υποστήρι, τη στήριξη με, νέων, με νέες πιστώσεις, θα μπορέσουμε να διαθέσουμε ε, και δύο-τρεις συνεργάτες στους, στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Εμείς πιστεύουμε, εάν οι συνεργάτες μας, και έχουμε πολλούς νέους εξαιρετικής ποιότητος συνεργάτες, εάν μπορούν να χειριστούν αυτά τα δύσκολα θέματα της οικονομικής απάτης, θα έχουμε και μεγαλύτερες ε, ε, επιτυχίες. Η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας και ο αντιπρόεδρος και που είναι και υπουργό Εσωτερικών είναι ο συνομιλητής μας. Εγώ συνάντησα τον Πρωθυπουργό δύο φορές, μιλήσαμε εις βάθος πάνω από μια ώρα ε, και τις δύο φορές για τα προβλήματα, είπαμε, εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας, τα προβλήματά μας ε, από την δικιά μας πλευρά, η πορεία που, που ακολουθεί η χώρα είναι, είναι σωστή, είναι καλή. Έχουμε ακόμα προβλήματα στη δικαιοσύνη. Τα προβλήματα στη δικαιοσύνη παραμένουν και ε, εγώ δεν πρόκειται μόνο το να ε, θέτουμε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων και να λέμε να η διαφθορά. Πρόκειται και, και για γνώση, ενημέρωση, ε, δυνατότητα πρόληψης και δυνατότητα επισήμανσης ε, μιας στραβοτιμονιάς, μιας υπόθεσης η οποία θα εξελιχθεί σε απάτη κλπ. Η γνώση λοιπόν, γνώση, εκπαίδευση, χρειαζόμαστε πόρους επαρκής για να μπορέσουμε να κλείσουμε και τις υποθέσεις αυτές. Τι νόημα έχει να συλλαμβάνονται ορισμένα άτομα και μετά να μένει ο φάκελος αυτός να μην κλείνει, να μην ολοκληρώνεται η υπόθεση. Ο πρώην Υπουργό δικαιοσύνη της Ρουμανίας είναι και εδώ τώρα μέλο του σώματο, και μπορεί ο ίδιος να σα πει πόσο δύσκολη είναι οι αλλαγέ στη δικαιοσύνη διότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και ιδίω στον τομέα της δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά δύσκολη η επιβολή αλλαγών. Άρα χρειάζεται και πίεση και ενίσχυση των γνώσεων δεν είναι μόνο τα λεφτά τα οποία μπορούν να λύσουν το θέμα, αλλά χρειάζεται και πρακτικη πρακτική μετάδοση γνώσεων, ένα πρακτικό know-how, να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές και πιστεύω ότι το κάνουμε αυτό. Και η συνεργασία μας εξελίσσεται καλά, θετικά. Όσον αφορά τώρα τα κτίρια, είχαμε κάνει μια ανακοίνωση τύπου, η οποία καταρχάς αφορούσε την πτέρυγα Σπινέλη Τέλος πάντων, πού βρίσκεται, μπροστά ή πίσω μας, το κτίριο Σπινέλη. Τη, τη δεκαετία του 90 είχε ε, προκύψει αυτό το πρόβλημα και είχε γίνει μια καταγγελία το 2001 για το κτίριο αυτό το εξετάσαμε, είχαμε εξετάσει τους ε, διαγωνισμούς που έγιναν, ε, δημοπρασίες, κατευθυντήριες γραμμές, προδιαγραφές κλπ μεγάλης δυσκολίας ε, δικαστικό ε, θέμα, νομικό θέμα. Ο διαμεσολαβητής, ε, πιστεύοντας ότι είμαστε και δικαστήριο εμείς, ε, μας ζήτησε να εμβαθύνουμε στη μελέτη αυτή, της καταγγελίας. Συζητήσαμε λοιπόν με τον διαμεσολαβητή, ε, κοιτάξαμε το φάκελο και θα το επενεξετάσουμε και με, το νομικό, με τη νομική υπηρεσία και θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, θα φέρουμε και τη νέα μας αξιολόγηση, τη νέα μας έκθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα από τα πιο δύσκολα και καυτά, είναι το πιο δύσκολο και καυτό θέμα που έχουμε ποτέ χειριστεί. Είναι ένα θέμα με νομικές διαστάσεις, ε, αν έχουν ερμηνευτεί σωστά οι διατάξεις του μειοδοτικού διαγωνισμού κλπ. κλπ. Για αυτά τα δύο κτίρια λοιπόν, μάθαμε μόλις τώρα ότι ο διαμεσολαβητής έχει διαπιστώσει τα ίδια προβλήματα, όπως είχαμε τότε με το Σπινέλη, και ότι έχει ζητήσει να γίνει μία έρευνα και σε αυτή τη στιγμή ε, είμαστε σε επαφή με τον διαμεσολαβητή, για, θα του στείλουμε μία επιστολή, να ρωτήσουμε τι στοιχεία έχει. Εμείς δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει καμία έρευνα, διότι όταν μας ήρθαν οι πρώτες ενδείξεις καταγγελίας, τα κτίρια αυτά δεν είχαν ακόμα ολοκληρωθεί. Τώρα λοιπόν πρέπει να, να γράψουμε στον διαμεσολαβητή και να του πούμε πέστε μας από πού να ξεκινήσουμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες υποψίες που έχετε ή καταγγελίες. Ο κύριος Έκανα λάθο, ε. Μου δώσαν λάθος όνομα. Δεν φταίω εγώ, όμως. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσει. αλλά θα πρέπει να φύγω αμέσως μετά για να ψηφίσω τον κύριο Βέρνερ Λάγκεν και θα στεναχωρηθεί αν δεν είμαι παρούσα στην ε, ε, ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει θα, μου, θα με ενημερώσουν για την απάντησή σας. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά τις αρμοδιότητές σας. Είπατε ότι δεν είσαστε δικαστική αρχή, ότι έχετε περιορισμό των αρμοδιοτήτων σας κλπ. Ε, αυτό, επειδή εγώ είμαι καινούριο μέλος, το ερμηνεύω σαν ε, να παραπονιέστε ότι οι αρμοδιότητες σας, το πεδίο αρμοδιοτήτων σας δεν αρκεί για να κάνετε καλά τη δουλειά σας. Ε, αυτό προσπαθείτε να μας πείτε Μήπως αν αυτό θέλετε να πείτε πρέπει να επαναξετάσουμε του χρόνου το θέμα των αρμοδιοτήτων, πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, αν δεν είσαστε ικανοποιημένοι. Και δεύτερον, στην έκθεσή σας γράφετε τις επιτυχίες που σημειώσατε για το λαθρεμπόριο τσιγάρων, την ε, διαφθορά στον αγροτικό τομέα και την παραχάριξη χαρτονομισμάτων. Ε, εμείς ε, τώρα σε πολλές επιτροπές έχουμε να συζητήσουμε το θέμα των, ε, των παρανόμων φαρμάκων, δηλαδή πιστεύετε ότι τα φάρμακα αυτά, τα παράνομα τα οποία κατασκευάζονται ε, είναι μια νέα αγορά η οποία έχει δημιουργηθεί, τα λιωμένα φάρμακα οι απομιμήσεις δηλαδή φαρμάκων και ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό στο μέλλον. Ο κύριο Μπρίνερ. Όχι, εγώ είμαι ευχαριστομένος με τις αρμοδιότητες που έχω. Δεν λέω. Τουλάχιστον με τις αρμοδιότητες οι οποίες προσδιορίζονται γενικά για το Όλαφ, έτσι. Για το γενικό πλαίσιο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να γίνουμε εμείς μία, ένας οργανισμός δίωξης ε, και επιβολής ε, ή ποινικών ερευνών. Όμως αυτό που θέλω είναι να μπορούμε να συνεργαστούμε με όλες τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που ξεκινάμε μία έρευνα αλλά γενικά, στη λεπτομέρεια δηλαδή υπάρχουν ορισμένα προσκόμματα. Γενικά όμως είμαστε ευχαριστημένοι με τις αρμοδιότητες. Όσον αφορά τώρα τα πλαστά φάρμακα, τις απομιμήσεις φαρμάκων, δεν είμαστε αρμόδιοι. Όχι ότι όταν διαπιστώσουμε ότι κυκλοφορούν πλαστά φάρμακα στην αγορά θα κλείσουμε τα μάτια. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να κινητοποιήσουμε το βιομηχανικό τομέα, τον παρασκευαστικό τομέα και να το σπίσουμε να συνεργάζονται πιο στενά μαζί μας για να ανταλλάξουν, να μας ενημερώνουν, να μεταδίδουν τις γνώσεις τους και όχι να ε, ε, κινούνται, να ε, ενεργούν σε στεγανά και να μην μας μεταδίδουν αυτά που ξέρουν για να μπορέσουμε και εμείς να ξεκινήσουμε τις έρευνές μας. Δεν, δεν υπάρχει πρόσκομα στο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με, τις παρασκευαστικές, με, τις, με τους παρασκευαστές. Δεν ζητάμε εμείς να μας ανακοινώσουν τα μυστικά ή να μας αποκαλύψουν ε, θέματα εμπιστευτικότητας. Εάν υπάρχει κάποια απάτη, μπορούμε να εξετάσουμε τις πτυχές, τις οικονομικές και άλλες, αλλά σαφή αρμοδιότητα, σαφή αρμοδιότητα για τα φάρμακα δεν έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της έκθεσης. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία φορά στις δημόσιες προμήθειες και την απάτη. Από τη δική μου την πείρα της καταπολέμησης της διαφοράς, οι, οι δημόσιες δαπάνες, οι δημόσιες προμήθειες είναι ε, από τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στον υψηλότερο σημείο για τη διαφθορά και ξέρουμε ότι γίνονται και δαπάνες ε, στα κράτη-μέλη μέσω κρατικών προμηθειών. Από τη δική σας την πείρα λοιπόν στην Όλαφ μπορέσατε να βρείτε κάποιο ε, πρότυπο απάτης μέσω ε, κρατικών προμηθειών, κάποιο μοντέλο απάτης. Αν η απάντηση είναι ναι, φυσικά θα μπορέσαμε να συνεργαστούμε και ε, ο στόχος μας θα είναι να ε, βρούμε έναν τρόπο να το μεταφράσουμε σε κανόνες αυτό. Επίσης, ε, τα σημεία επαφής της Όλαφ με τους εθνικούς εταίρους. Όπως είπατε και εσείς μόνο σας, η δουλειά της Όλαφ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα εθνικά σημεία επαφής. Πώς τα αξιολογείτε, πώς αξιολογείτε τη δουλειά τους, θεωρείτε ότι υπάρχουν κοινά κριτήρια που ισχύουν για όλους. Και μια δεύτερη ερώτηση. Υπήρχαν περιπτώσεις ε, στις οποίες υπήρχαν πληροφορίες ή λόγοι που σας έκαναν να αφισβητήσετε την ακεραιότητα των ανθρώπων που εργάζονται στα εθνικά σημεία επαφής. Και αν ναι, τι κάνατε σε αυτή την περίπτωση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στο τελευταίο σκέλος της ερώτησης, δηλαδή σε επαφές που έχουμε με τα νέα κράτη-μέλη μέσα στο πλαίσιο ΑΦΚΟΣ, δηλαδή έτσι ονομάζεται η συντονιστική αυτή δράση επαφών. Δεν μπορώ να κάνω μία ισοποδετική κριτική και να κρίνω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Βασίζουμε τη συνεργασία μας σε ορισμένα ουσιώδη θέματα. Και όπως σας είπα, συνεργασία με αυτούς ε, τους ανθρώπους, με τα στελέχη επαφής δηλαδή, εξελίσσεται θετικά προς την σωστή κατεύθυνση. πολλές φορές όταν ε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα επιτύχαμε να επιβάλλουμε μία αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για να στρώσει η κατάσταση. Ε, ε, ε, ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα μεμονωμένα σημεία επαφής, στους ανθρώπους ή φορείς και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα προς το παρόν, ούτε έχουμε διαπιστώσει ένα έλλειμμα ακιαρεότητος σε αυτές τις επαφές. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει και είμαι πολύ προσεκτικό στη διατύπωσή μου. Ε, υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μία κουλτούρα σε ορισμένα κράτη να κρατούν μυστικά τα μειονεκτήματά τους. Δηλαδή, ε, ότι, τα στραβά δεν θέλουν να τα βλέπει η δημοσιότητα, δεν θέλουν να προβάλλουν έξω προς τα έξω τα, τα σφάλματά τους, τις αδυναμίες τους και ότι πάει στραβά. Αυτή την κουλτούρα προσπαθούμε να την αλλάξουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίζουμε τα λάθη και να τα διορθώνουμε. Για τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Βεβαίως εκεί είναι ένα σημείο εντοπισμού πολλών, πολλών προβλημάτων. Πέραν των διαγωνισμών αυτών καθεαυτών, τα, τα περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονται στην εφαρμογή. Δηλαδή γίνεται η, η σύμβαση και μετά σημειώνονται, εντοπίζονται τα προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει στις προδιαγραφές των διαγωνισμών αυτών να, έχουμε ένα καλύτερο έλεγχο, μια καλύτερη εποπτεία των προδιαγραφών αυτών για να μπορέσουμε προληπτικά να δούμε, να εντοπίσουμε εάν ορισμένες προδιαγραφές, ορισμένα κριτήρια τα οποία τίθενται μέσα σε αυτούς τους μειοδυτικούς διαγωνισμούς είναι ευάλωτα ή οδηγούν ή επιτρέπουν παρανομίες και ατασταλίες και να τα προλάβουμε αυτά πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Είναι ένας τεράστιος τομέας αυτός με πολλές παγίδες. Ε, είμαι της γνώμης ότι στα νέα κράτη-μέλη ιδιαίτερα, αλλά και στην Κομισιόν, έχει σημειωθεί μια πολύ θετική εξέλιξη, ε, επειδή έχουν καταλάβει καλύτερα, έχουν συνειδητοποιήσει καλύτερα τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν οι απάτες. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι νέο μέλος της Επιτροπής. Ε, κατά συνέπεια θα με συγχωρήσετε για μερικές θεμελιώδεις ε, ερωτήσεις. Είπατε ότι εποφεληθήκαμε κατά 250 εκατομμύρια ευρώ από τις δραστηριότητες της Όλαφ σε σχέση με ένα προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια. Τώρα αυτό μπορεί να είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι ένδειξη αποτελεσματικότητας ή ένδειξη πολύ μεγάλης έκτασης ε, του φαινομένου της απάτης και της διαφθοράς. Τι από τα δύο είναι. Έχετε κάποια αίσθηση του μεγέθους του αντικειμένου που είναι στην αρμοδιότητά σας. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, μιλήσατε για κάποιες χώρες. Έχετε, θα μπορούσατε να μας πείτε, περιοχές υψηλού κινδύνου. Περιοχές δηλαδή ε, δραστηριότητας που θεωρείτε ότι εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα περισσότερο συχνά από ό,τι σε άλλες. Ευχαριστώ. möchte nur 450 Millionen. 450, 450 εισπράξαμε μεγάλο ποσό. Όχι ότι όλη η ζημιά ήταν τόση μόνη προς Θεού, αλλά ε, πρέπει να τονίσω ότι με τα πολλά μέτρα που εφαρμόσαμε, ό,τι δεκάρα μαζεύουμε, τη μαζεύουμε με πολύ δύσκολες συνθήκες, ό,τι ευρώ μάλλον. Και είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή, το τονίζω. Και όσοι βρίσκονται σε τρίτες χώρες ή σε άλλες χώρες, ξέρουν ε, πόσο δυναμικά επεμβαίνουμε όταν κάτι ε, πάει στραβά. Βεβαίω ορισμένα πράγματα θα στραβώσουν, δεν, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Ακόμα και στο πιο καλά οργανωμένο κράτος δημιουργούνται προβλήματα. Υπάρχουν ε, κράτη τα οποία ε, σέβονται το Διεθνή Κώδικα Διαφάνειας, όμως σε κάποια στιγμή παρουσιάζεται μία περίπτωση διαφθοράς. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και το ΟΛΑΦ και η Κομισιόν κάνουμε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και στον έλεγχο και στην ίσπραξη των ε, ποσών που, που πρέπει να επιστραφούν με ένα budget 50 εκατομμυρίων ε, είναι ζόρι, είναι, είναι, μικρό αυτό το budget, διότι εδώ μιλάμε για τεράστιες απάτες και οι λογαριασμοί, δηλαδή αυτά που ξοδεύουμε εμείς για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη ενός φακέλου, είναι πολύ ψηλοί. Εγώ σας ανέφερα ορισμένα στοιχεία, γιατί δεν θέλω να σας παρουσιάσω στατιστικά στοιχεία, γιατί είναι αδύναμα. Σας παρουσίασα απλώς ορισμένα ισχυρά στοιχεία για να δείτε την έκταση των δραστηριοτήτων μας. Εγώ δεν θέλω να κάνω, ε, να σας παρουσιάσω εικασίες ή αυθαίρετα ε, ε, στοιχεία. Πολλές φορές ε, θα μπορούσα εύκολα να σας πω ότι εξετάσαμε πέντε περιπτώσεις από 600 φακέλους που έχουμε στο γραφείο μας. Άρα λοιπόν έχουμε 600 ε, περιπτώσεις απάτης. Το να ε, σας δώσω τέτοια αυθαίρετα στοιχεία δεν είναι σωστό, διότι εγώ θέλω να σας μιλήσω για υποθέσεις που στηρίζονται σε συγκεκριμένες αποδείξεις, όχι σε ενδείξεις. Δεν ξέρω πόσο είναι συνολική ζημιά της οικονομικής απάτης, ούτε μπορώ να κάνω μια εκτίμηση έτσι ε, ε, ad hoc, ε, από το κεφάλι μου, από το μυαλό μου, αλλά τα 450 εκατομμύρια είναι ένα ποσό σοβαρό και, και αισιόδοξο, διότι δείχνει ότι ενεργούμε σωστά το ποσό αυτό της ίσπραξης ε, ε, μπορεί να μειωθεί τα επόμενα χρόνια, διότι έχουμε αυξήσει πάρα πολύ την πρόληψη των απατών ε, και των, της διαφθοράς. Εφόσον λοιπόν αυξάνεται η πρόληψη, μπορεί ενδέχεται να μειωθούν και τα ποσά που εισπράττουμε εν τέλει ή που επιστρέφονται τέλος πάντων. Και, και τι άλλο ρωτή... Ναι. Λοιπόν, Βεβαίως υπάρχουν περιοχές όπου ο έλεγχος είναι πολύ αποτελεσματικός και καλός στον γεωργικό τομέα. Γίνονται ενδελεχείς, ουσιώδης και εις βάθος έλεγχος με μετρήσιμα μέσα και έτσι έχει μειωθεί πάρα πολύ το ρίσκο ε, των απατών. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι να σημειωθούν απάτες, ιδίως στον τελωνιακό τομέα, ιδίως στα προτιμησιακά καθεστώτα, δηλαδή εκεί όπου μια χώρα έχει μια, ένα ειδικό προνομιακό καθεστώς για ε, τελωνιακές και δασμολογικές υποθέσεις, Εκεί μπορούν ακόμα να παρουσιαστούν υποθέσεις λάθρεμπορίας και υπάρχει αυτό το ρίσκο. Όμως, όταν μια χώρα είναι πολύ ακριβή, έχει ας πούμε ακριβές ε, τιμές, π.χ. ας πούμε στα τσιγάρα, εντάξει, ενδέχεται εκεί να σημειωθεί λαθρεμπόριο. Αλλά αυτό <laughs> τι να κάνουμε, δεν είναι δικό μα πρόβλημα η ακρίβεια ή όχι των κρατών. Και βέβαια υπάρχουν προγράμματα που είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Ας πούμε, στην ε, διαρκή ε, εκπαίδευση, κατάρτιση ε, ένα σεμινάριο, έτσι, διαρκούς εκπαίδευσης, κατάρτισης. Μας λένε ότι συμμετείχαν 150 άτομα. Ε, ήταν 150 ή ήταν 15. Ε, είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή των ελέγχων και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε ορισμένες αναφορές που μας δίνονται. Και για να έχουμε υποψίες, για να εξετάσουμε, να δώσουμε συνέχεια σε μία υποψία, πρέπει να έχουμε σαφείς ενδείξεις. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ορισμένοι φορείς ή οργανισμοί είναι, ε, χαίρονται που παίρνουν κονδύλια, παίρνουν επιστώσεις, μετά όμως δεν, δεν ξέρουν τον καλύτερο τρόπο να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ανταγκαστικά ότι κάνουν μια απάτη. Ενδέχεται να, να χρηματοδοτούν παλαιότερες δραστηριότητες, ενώ οι πιστώσεις αυτές τους έχουν δοθεί για την έναρξη καινούριων προγραμμάτων, χωρίς αναγκαστικά να υπάρχει μια σκόπιμη ε, παραπλάνηση. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι πολύ πολύ σημαντικά για μας και γι' αυτό θέλουμε να εφαρμόσουμε προληπτικά μέτρα. Ο κύριος Ανδρέας. Thank you, Mr. Chairman. Κυρία. Mr. Brunner, thank you for your Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπρούνερ, σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και ε, ευχαριστούμε και για την πρόσκληση στην Όλαφ για να δούμε πώς δουλεύετε. Εγώ σίγουρα θα έρθω. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι νέο μέλος του Κοινοβουλίου, αλλά δεν είμαι καινούρια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μπορεί να με αναγνωρίζετε κάποιοι από εσά. Και πρέπει να πω ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω τα στατιστικά σας στοιχεία, διότι δεν μπορώ να κατανοήσω τι σχέση έχει η αύξηση ή η μείωση ε, περιπτώσεων με την αύξηση ή τη μείωση των παρατυπιών ή την αύξηση ή τη μείωση της αποδοτικότητάς σας και του τρόπου που διεξάγετε τις εργασίες σας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι σας οδηγεί στο άνοιγμα μιας υπόθεσης ώστε να μπορέσω να κατανοήσω λίγο και τα στατιστικά σας στοιχεία. Και μια δεύτερη ερώτηση είναι ότι είπατε ότι είστε εντελώς ανεξάρτητοι. Εξ όσων γνωρίζω, ε, είστε υπόλογοι στον Επίτροπο Υπεύθυνο για τον Προϋπολογισμό. Πού ακριβώς έγκυται λοιπόν η ανεξαρτησία σας. Ευχαριστώ. για να είμαι σαφής. Εγώ παρουσιάζω την έκθεσή μου στο Κοινοβούλιο, είμαι υπόλογος στο ή μάλλον όταν με καλεί το κοινοβούλιο παρουσιάζω την έκθεσή μου στη δημοσιότητα με διαφάνεια και την ίδια διαδικασία εφαρμόζουμε και στην Κομισιόν όπου συζητούμε εσωτερικές υποθέσεις. Αυτή είναι η μόνη γραμμή αναφορά στην οποία έχουμε. Αυτά τα οποία παρουσιάζω στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προστατεύονται γενικώ από την διαδικασία του, χειρισμού των πληροφοριών ε, αλλά δεν υπάρχει καμία, κανένας περιορισμός στο τι θα παρουσιάσω, τι θα αναφέρω. Ε, αυτή την έκθεση παρουσιάζει ο διευθυντής του Όλαφ στα θεσμικά όργανα. Ε, τώρα πώς ξεκινάμε μία υπόθεση, δεν θα πάω εγώ σε έναν επίτροπο και θα του πω «Μου επιτρέπετε κύριε επίτροπε να ανοίξω αυτό το φάκελο ή όχι». Γι' αυτό ακριβώς παλιότερα είχαμε τονίσει την επισημία μας να είμαστε ανεξάρτητο όργανο έναντι των θεσμικών οργάνων και ε, ε, είχαμε επικρίνει τις προτάσεις της κομισιό παλιότερα βεβαίως που δεν είχε σεβαστεί την αντικειμενικότητα του Όλαφ. Από τότε μέχρι τώρα ποτέ Ποτέ δεν μου είπε κάποια αρχή ισότιμη ή προϊσταμένη αρχή ε, τι να φάκελο να ξεκινήσω, ούτε επηρεάστηκα ποτέ, ούτε υπήρχε οποιαδήποτε επιρροή από άλλο φορέα ή όργανο προς εμάς να, να ανοίξουμε, να κλείσουμε κάποιο φάκελο. Εμείς ενεργούμε ανεξάρτητα προς όφελος του οργανισμού μας, της υπηρεσία μας. Είναι προφανές ότι εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε βασικά τους στόχους του δικού μας οργανισμού. Ε, δεν ε, ανοίγουμε φακέλους έτσι αυθαίρετα ή επειδή μας αρέσει, ούτε ξεκινάμε ε, φακέλους εναντίον κάποιου ατόμου επειδή δεν μας αρέσει υπάρχει μια υποκειμενική κρίση αλλά ο στόχος μας είναι γνώση του του παρελθόντος, δηλαδή τα παθήματα μαθήματα, εννοούμε παθήματα υποθέσεων, τι γνώσεις μπορούμε να κερδίσουμε από παλιές υποθέσεις και συμβάντα που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε και να ανοίξουμε μελλοντικού φακέλους. Εγώ στις δραστηριότητε μου είμαι απόλυτα αντικειμενικός και ανεξάρτητος και όλοι το έχουν σεβαστεί μέχρι τώρα. Τώρα μου λέτε τι στοιχεία χρειάζεται το όλα για να ξεκινήσει μια υπόθεση. Θα σας παρακαλούσα να ε, μελετήσετε τις εκθέσεις τις οποίες έχουμε υποβάλει κατά το διάστημα αυτό των ετών και να μελετήσετε ε, την εντολή την οποία έχουμε λάβει, η οποία εντολή από τα θεσμικά όργανα ε, αναφέρει σαφέστατα πότε, πώς και γιατί ανοίγει ένας φάκελος. Ένα φάκελο, μια υπόθεση ανοίγει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά μας έχουν δοθεί, ήταν μέρος της εντολής μας, βάσει του κανονισμού σύστασης του Όλαφ και αυτές τις κατευθυντήριες γραμμέ ακολουθούμε. Τώρα, ο έλεγχο των δραστηριοτήτων μας ε, ε, έχει αντιγραφεί και από άλλου διεθνεί οργανισμού. Η φάκελη διαχείριση των υποθέσεων μας αποφασίζεται σε μια 100% διαφανή διαδικασία του εκτελεστικού συμβουλίου, του διοικητικού οργάνου του Όλαφ, το οποίο πρέπει να δικαιολογήσει γιατί και πώς άνοιξαν οι φάκελοι, ποιες υποθέσεις. Βεβαίως εγώ υπογράφω τις αποφάσεις, αλλά Πίσω μου έχω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο με καλύπτει στις αποφάσεις αυτές. Και αυτή είναι και η εγγύηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας μας, η κυρία Γκρέσλα. Ευχαριστώ τον κύριο ε, Μπρούνο και Μπρίνερ και την, την, το Όλαφ, την Σας συγχαίρω για τα 10 χρόνια που γιορτάζετε. Πιστεύουμε ότι το Όλαφ είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο έγινε αν και έχει λίγο αδρανήσει, όχι αδρανήσει, αλλά έχει πέσει λίγο ο ενθουσιασμός τελευταία. 130 τροπολογίες για το Όλαφ έχουμε αποφασίσει και το Νοέμβριο στο Σώμα, στο Κοινοβούλιο, αποφασίσαμε και την, νομική, την νέα νομική βάση. Ε, είσαστε ικανοποιημένοι με αυτές τις αποφάσεις του περσινού Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Κομισιόν είπατε ε, και σωστά είπε και ο κύριος Μπαρόσο ότι το Όλαφ πρέπει να είναι εντελώ ανεξάρτητο, ότι ε, η παλιότερη έκθεση λοιπόν για το Όλαφ έχει εκπέσει, δεν ισχύει πλέον ή δεν ήταν ανεξάρτητο το Όλαφ παλιά. Τι σημαίνει τώρα πλήρης ανεξαρτησία, ήταν εν μέρη ανεξαρτησία στο παρελθόν. Τώρα, ε, εφόσον λοιπόν ο, νέος, ο πρόεδρος της Νέας Επιτροπής ζητάει πλήρη ανεξαρτησία, τι εννοεί καλύπτει και της, ε, την προστασία δεδομένων. Με τη νέα πρόταση υπάρχει ο κίνδυνος το Όλαφ να δραστηριοποιείται σε υποθέσεις μόνο κατόπιν εντολής της ε, Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό, διότι μέχρι τότε δεν ήταν έτσι, άρα πρέπει να καταψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε, στην έκθεση αυτή του Προέδρου της Επιτροπής αναφέρονται και θέματα για την προστασία δεδομένων, νέα στοιχεία δηλαδή. Συμφωνείτε με αυτά, διαφωνείτε, πώς κρίνετε αυτή την έκθεση των νέων δραστηριοτήτων. Έχω και μια τρίτη ερώτηση. Έγινε μια έρευνα για την εσωτερική έκθεση του Κοινοβουλίου για τη χρήση πιστώσεων κονδυλίων μέσω συναδέλφων και εν συνεχεία επικράτησε σιωπή. Πόσες υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις εθνικές δικαστικές αρχές, τι αφορούν και πότε θα μάθουμε, θα ενημερωθούμε το τι έγινε σε αυτές τις υποθέσεις, διότι πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζημιώθηκαν σημαντικότατα από την έκθεση αυτή. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, εφόσον υπήρξε ένα κατηγορητήριο, τι έγινε με αυτό. Ορισμένες φορές ε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ενημερωνόμαστε σωστά και έγκαιρα, ε, αλλά μερικές ε, φορές ενημερωνόμαστε από το ίντερνετ. Σε μία περίπτωση της Βουλγαρίας, μία λεγόμενη ομάδα Stoikov ας πούμε, ανακοίνωσε στις βουλγαρικές αρχές 50 περιπτώσεις απατών που είχαν σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Μέσω του, των ιστοσελίδων ε, λοιπόν ενημερωθήκαμε και θα θέλαμε να ξέρουμε αυτές 50 περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν στο ίντερνετ, τι έγινε με αυτές. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μπρίνερ, εγώ είπα ότι είμαι ικανοποιημένος, αλλά αυτά όλα εξαρτώνται από τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες μας. με τις χώρες αυτές, τις προβληματικές που ανέφερα. Ε, Βεβαίω υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωση τη συνεργασία. Λέω ότι είμαι ικανοποιημένο ε, με την πορεία που ακολουθείτε. Ε, οι διαδικασίες τώρα που αφορούν μέλη του σώματος, τωρινά ή προηγούμενα, παρελθόντα, μέλη, τι έγινε με αυτές τις υποθέσεις. Ε, ε, θετικό αποτέλεσμα είχαμε, κυρία Γκρέσλε. Εγώ δεν θέλω να δακτυλοδεικτώ κάποιον, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να το κάνω αυτό έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε λάβει μια έκθεση τότε με εκατοντάδες ονόματα προς εξέταση και ήταν σαφές ότι μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία ένας πολύ μικρός αριθμός ε, ευρωβουλευτών άξιζε, έπρεπε να εξεταστεί ουσιαστικά ε, πριν υποβάλλουμε μια ελεγκτική έκθεση πρέπει να εφαρμόσουμε πολύ σωστά όλες τις διαδικασίες, να κάνουμε όλες τις έρευνες που χρειάζονται και έτσι ο ρυθμός από όλες αυτές τις, από τη λίστα αυτή την τεράστια των ευρωβουλευτών που μας ήρθε και τελικά ο ρυθμός των ευρωβουλευτών που παρανόμησαν ή παραβίασαν κανονισμούς είναι μικρός. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τον έλεγχο ορισμένων μελών, ξεκινήσαμε ορισμένες υποθέσεις, μικρός αριθμός δηλαδή. Ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας ε, βοηθήσει με τα αναγκαία στοιχεία που χρειάζεται για την ε, μελέτη των φακέλων. Εν συνεχεία έγιναν οι εκλογές ε, του Κοινοβουλίου, φύγαν μέλη, ήρθαν καινούρια. Και όπως σας είπα, εγώ δεν μπορώ να κατονομάσω, ούτε θέλω να κατονομάζω υπόπτους, αλλά έχουν ξεκινήσει, έχουν ανοίξει ορισμένοι φάκελοι. Μου, μου είχατε ζητήσει τότε παλιότερα να ολοκληρώσουμε τους φακέλους αυτούς, να τους κλείσουμε την άνοιξη φέτος, πριν από τις εκλογές. Αλλά δυστυχώς ούτε καν είχε ξεκινήσει η ουσιαστική δουλειά δεν μπορούμε, μπορέσαμε σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα να ξεκινήσουμε και να ερευνήσουμε όλες τις, τα ονόματα αυτά που μας είπαν. Και να ερευνήσουμε κάθε καταγγελία και κάθε λεπτομέρεια του φακέλου. Επίσης είχαμε και προσκόμματα από πλευράς ε, μελών ή κοινοβουλίου. Δεν μπορέσαμε να έχουμε τα, στοιχεία που θέλαμε εγκαίρως, διότι καταλαβαίνετε υπήρχαν ορισμένε αντιδράσεις. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ε, λείπει μια συνολική αξιολόγηση του φακέλου, λείπουν ακόμα στοιχεία που θα μας διευκολύνουν να κρίνουμε την υπόθεση και υπάρχουν και κρεμείς δικαστικές υποθέσεις που, δεν έχει βγει ακόμα απόφαση. Θα εργαστούμε με, κάθε, με όλες μας τις δυνάμεις να ολοκληρώσουμε αυτές τις υποθέσεις δεδομένου ότι αφορούν μέλη του σώματος, νυν και παρελθόντα και ιδίως και επανέρχομαι στο θέμα της Βουλγαρίας που μας καίει, σαφώς όλοι αναγνωρίζουμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε πολλά πρέπει να κάνουμε, ε, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και δεν μπορούμε έτσι από σήμερα σε αύριο να επιβάλλουμε αλλαγές σε ένα σύστημα δικαιοσύνης, σε, μια χώρα. Α, και ξέχασα να απαντήσω και σε ένα άλλο σκέλος, η μεταρρύθμιση του Όλαφ. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν έκανε μία δήλωση πολιτικής φύσεως, την οποία ερμονεύω ως εξής ότι δεν θα ξεκινήσουμε εμείς φτού και από την αρχή με ένα νέο οργανόγραμμα ή ένα νέο σχέδιο λειτουργίας λόγω της ε, ε, αναθεώρησης που υπάρχει ακόμα στο, στο τραπέζι μας. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε με την πορεία που ακολουθήσαμε και παλιότερα με ορισμένες ίσως αλλαγές. Δηλαδή, οποιαδήποτε αλλαγή επέλση θα είναι προς το προς όφελός μας ε, για να λειτουργούμε καλύτερα. Ε, θα πρέπει να εξεταστούν και νομικές επιπτώσεις βεβαίως, η νομική βάση των μεταρρυθμίσεων και πιστεύω ότι οι δηλώσεις αυτές ε, του Προέδρου της ε, Κομισιόν ε, δείχνουν ότι έχουμε λειτουργήσει σωστά, έχουμε δουλέψει σωστά μέχρι τώρα και ότι όλα τα μέτρα τα οποία τυχόν θα εφαρμοστούν τα καινούργια στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση του οργανισμού μας και όχι στην οπισθοδρόμηση ε, περαιτέρω εξέλιξη λοιπόν, όχι νέα οργάνωση. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του, τον εκπρόσωπο της Όλαφ. Όπως ξέρετε έχουμε νέα θητεία, υπάρχουν και νέες φυσιογνωμίες και παλιές φυσιογνωμίες, οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η πρώτη επαφή. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, όχι μόνο για να ενημερωθώ εγώ, αλλά και για να είναι ενήμερα και τα μέλη της Επιτροπής μας, Ιστορικά έχουμε το κώδικα διοντολογίας για άτομα τα οποία ε, έχουν ε, ε, συμφέροντα. Υπάρχει και ο επιθεωρητής, ε, ο οποίος εξετάζει τα θέματα στο οργανόγραμμα της Όλαφ. Θα ήθελα να μας κάνετε μια μικρή περιγραφή για το πώς λειτουργεί το σύστημα, αν λειτουργεί και αν υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μπορείτε να μας παρουσιάσετε για να μας πείτε αν είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο και ίσως θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τη βελτίωσή του. Θα θέλαμε επίσης να μας σχολιάσετε λίγο καλύτερα το θέμα της σχέσης ε, με την Επιτροπή ε, Εποπτείας της Όλαφ. Η εποπτεία, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντική δουλειά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει να κάνει και με τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της Όλαφ για να μπορέσει να προχωρήσει και με τα καθήκοντά της. Θα ήθελα να τα ξέρω αυτά λίγο για να είναι ενημέροι όλοι οι συνάδελφοι, αλλά και γιατί υπάρχει μια νέα ε, κατάσταση σε αυτή τη νέα θητεία. Επομένως θα πρέπει να μας πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτός ο οργανισμός υποπτία. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε τι συμβουλέ ή τι συστάσεις θα δίνατε ώστε διότι κάθε φορά πηγαίνουμε στις χώρες μας δεν έχουμε ακριβώ επικρίσει, αλλά Θέλουν να γνωρίζουν. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η δουλειά τη Όλαφ και περνάει από εκεί και πέρα η υπόθεση με όλα τα στοιχεία σε ένα κράτο μέλο. Πώς παρακολουθείτε εσείς τι γίνεται από εκεί και πέρα από πλευρά Όλαφ και πώς μπορεί να ε, προχωρήσει αυτή η παρακολούθηση. Χάνεται, κόβεται το νήμα ή μπορούμε να έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Και τέλος, σήμερα το, φέτος το καλοκαίρι στον τύπο είδαμε κάτι που εμένα μου φάνηκε ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ήταν ένα σχόλιο που αφορούσε στο Γαλιλαίο και το πώς αποφασίστηκε και εφαρμόστηκε η χρηματοδότηση του Γαλιλαίου που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχει ειδικό ενδιαφέρον και αυτές οι πρωτοβουλίες είναι που βοηθούν την Ευρώπη να προχωρήσει ως χώρος ε, καινοτομία και τεχνολογίας. Θα ήθελα να ξέρω εάν η Όλαφ λοιπόν έχει λάβει κάποια ενημέρωση για αυτές τις επικρίσεις από πλευρά εσωτερικών ελεγκτών ε, για τη χρηματοδότηση του Γαλιλαίου. Ευχαριστώ. Äh, Αν σας κατάλαβα καλά, αναφέρεστε σε εσωτερικού κανονισμούς. Έχουμε το εγχειρίδιο, το καταστατικό λειτουργία μας, το οποίο το εξυγχρονίζουμε τώρα και πολλές αλλαγές τις οποίες θα έχει θα καλύπτουν και τη διαδικασία εσωτερικής εποπτείας, εσωτερικού ελέγχου. και άλλες ε, αλλαγές ε, κατόπιν συστάσεων της Κομισιόν. Γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή μία αναθεώρηση του καταστατικού λειτουργίας μας και με διαφανή τρόπο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η... το καταστατικό μας έχει αντιγραφεί και από άλλους οργανισμούς που θέλουν να λειτουργήσουν βάσει των δικών μας προτύπων. Τώρα, τι γίνεται με τη δικαστική εξέλιξη υποθέσεων ε, τις οποίες έχουμε χειριστεί εμείς και προωθήσει σε εθνικές αρχές, ε, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Φανταστείτε τι χρόνο και χρήμα θα χρειαζόμαστε να παρακολουθήσουμε και τους φακέλους όλους αυτούς αφού τους προωθήσουμε εμείς. Ήδη εμείς ε, δαπανούμε χρόνο και χρήμα για τη μελέτη των δικών μας φακέλων στα δικά μας γραφεία. Λοιπόν, υπάρχουν φάκελοι, τους οποίους έχουμε στείλει. Παραδείγματο χάρη στην Ισπανία υπάρχει μία υπόθεση, η οποία κράτησε εννέα χρόνια. Εννέα χρόνια ήταν υπόθεση αστικού δικαίου και έκλεισε φέτος, μετά από εννέα χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι... Τι χρόνος χρειάζεται και τι δικαστικός ε, λαβύρινθος ανοίγεται ε, η Όλαφ επιμένει βεβαίως, εάν είναι οικονομική απάτη, να πάρει πίσω τα χρήματα. Έτσι. Μία φορά είχαμε ανοίξει μία, ένα ποινικό φάκελο, το στείλαμε στο αρμόδιο κράτος μέλος, το κράτος μέλος μας είπε ε, τρίχες, δεν είναι σωστή αυτή η υπόθεση, όμως εμείς επιμείναμε και τελικά πάλι μετά από χρόνια καταφέραμε και εισπράξαμε τα χρωστούμενα. Έχουμε ε, καθίσαμε δηλαδή με, για την υπόθεση αυτή μαζί με την Κομισιόν και είπαμε αυτά τα χρήματα ντε και σόνι πρέπει να επιστραφούν. Και το καταφέραμε παρόλες τις αντιρρήσεις της δικαστικής αρχής. Πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μας δικαίωσε και τελικά μετά από 9 χρόνια επιτέλους εισπράξαμε αυτά τα λεφτά. Ε, ναι, δεν είναι εύκολο να πείσουμε κάποιον που καίγεται για να δει τα αποτελέσματα μιας υπόθεσης ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος να κλείσει ένα φάκελο Ομολογώ ότι δεν είναι ικανοποιητική αυτή η κατάσταση, αλλά δεν είναι και στα χέρια μας. Και στο Βέλγιο, και στο Βέλγιο έχουμε ακούσει πάρα πολλά ε, παράπονα. Έχω ακούσει χιλιάδες παράπονα και από πλευράς Βελγίου ε, για την αργή διεκπαιρέωση των υποθέσεων, τι να κάνουμε, το συζητούμε όλα αυτά συνεχώς. Είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τέτοιες περίπλοκες διαδικασίες. Δεν είναι μόνο περίπλοκες στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δι Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και στο εθνικό επίπεδο. Προσπαθούμε πάντως. Η εσωτερική εποπτεία του οργανισμού μας δεν έχω να πω τίποτα. Έχουμε ένα νέο ε, Έχουμε έναν ε, νέο άτομο επικεφαλής της γραμματείας, ε, σύμβουλο, τον οποίο ανέλαβε τη θέση του τα, τις, τελευταίες, τις πρόσφατα, τις τελευταίες μέρες και η τελευταία επιτροπή εποπτείας ανανέωσε τη δεύτερη εντολή. Έχουμε την Επιτροπή Εποπτείας, η οποία λειτουργεί πλήρως. Θα δούμε τώρα στο μέλλον πώς θα λειτουργήσει, πώς θα εξελιχθεί αυτή η εποπτεία εσωτερική. Δεν ε, συμμετέχω εγώ, αλλά είναι η υποπτική μου αρχή η οποία καθορίζει και τη διαδικασία εποπτείας και τους μηχανισμούς εφαρμογής δεν είμαι εγώ σε θέση να αποφασίσω πώς θα κάνω εγώ τον εσωτερικό μου έλεγχο. Και επαναλαμβάνω, εάν πει κάποιος, ε, μας κατηγορήσει ότι εδώ ας πούμε η χρηματοδότηση είναι, δεν είναι, είναι αδιαφανής ή δεν μ' αρέσει αυτό το οποίο γίνεται, ε, ή μας ε, πει ότι εδώ υπάρχει κάποια χειραγώ... κάτι δεν πάει καλά, κάτι εδώ είναι στραβό. Αν κάποιος μας κάνει μια καταγγελία τέτοιας φύσεως, ε, ε, δεν αρκεί να ξεκινήσω μια υπόθεση με υποψίες. Πρέπει να έχω συγκεκριμένες ενδείξεις, στοιχεία δηλαδή, βάσιμα. μία πολιτική γκρίνια ή μία πολιτική δυσαρέσκεια δεν μου φτάνει για να ξεκινήσω εγώ μία υπόθεση. Δώστε μου αυτά στοιχεία και είμαι εντάξει. Κύριε Μπρούν, Μπρούνερ, ας ε, κλείσω εγώ με κάποιες ερωτήσεις, μια και δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα κάνω τι τελευταίε λοιπόν, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις και στι 4.30 πρέπει να τελειώσουμε τη συνεδρίαση. Τα, ερωτήματα θα είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι απλός όσο μπορώ. Καταρχάς, ε, ποια είναι η κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της ΟΛΑΦ και των εθνικών δικαστικών αρχών στις διάφορες χώρες. Ποια είναι η σχέση των μεν με τους δε. Υπάρχουν ποινικέ δίκες που είναι πολύ μακρές, τραβανείς μάκρο σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζομαστε χρόνια για να φτάσουμε σε καταδίκες. Η Όλαφ παρόλα αυτά είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει κάποια ερευνητικά στοιχεία που προκύπτουν από διάφορες έρευνες των εθνικών ε, ερευνητικών αρχών. Κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητα από την τελική ας πούμε, έκβαση της ε, διαδικασίας, της ποινική διαδικασίας. Επίσης, τι προστασία, τι κυδαιμονία μπορεί να παράσχει η, η Όλαφ στους πληροφοριοδότες που της δίνουν βάσιμα στοιχεία. Και το τελευταίο στοιχείο. Νομίζω Κάπως την κάλυψε ένα συνάδελφος. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι τι γίνεται με τις ε, παραβιάσεις ε, στους διαγωνισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη νομοθεσία. Η νομοθεσία αυτή γίνεται σεβαστή. Και τελικά τι κάνει όλα, τι προτίθεται να κάνει για να επαληθεύσει την ε, νομοτυπία των διαγωνισμών αλλά και την εκτέλεση των έργων. Εγώ ασχολήθηκα επί χρόνια με τέτοια, με τέτοια θέματα και ξέρω πολύ καλά ότι οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις είναι ο βασικός τομέας όπου υπάρχει συμπεγνία μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και πολιτικών φορέων. Εδώ δηλαδή είναι ο πυρήνας της διαφθοράς. Σκοπεύει όλα αυτά τα επόμενα χρόνια να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, δηλαδή μέσω των δημοσίων ε, χρηματοδοτήσεων, μέσω της διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων αυτών, μπορεί να σταματήσει αυτή την διάβρωση των θεσμών από το οργανωμένο έγκλημα. Μπορεί, ας πούμε, να κάνει κάτι όλο για αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ε, äh, Η συνεργασία με τις δικαστικές αρχές έτσι όπως ε, την κρίνουμε εμείς, εθνικές εννοώ δικαστικές αρχές, λειτουργεί θαυμάσια διότι έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο μεταξύ του Όλαφ και των εθνικών δικαστικών αρχών. Δηλαδή, δεν λέμε ότι οι δικαστικοί λειτουργοί αντιτίθενται ή δεν θέλουν να χειριστούν αυτούς τους φακέλους αλλά ε, εξαρτάται και από τα συστήματα του δικαίου που ισχύουν σε κράτες, στα κράτη-μέλη. Πολλοί φάκελοι, αντί να είναι πάνω-πάνω, στα γραφεία των δικαστικών λειτουργών είναι από κάτω. Εξαρτάται τι προτεραιότητες υπάρχουν, ε, τι φόρτος εργασίας υπάρχει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η διάσκεψη των εισαγγελικών αρχών στη Βιέννη όπου ε, θα συγκεντρωθούν όλοι οι εισαγγελείς των κρατών μελών που είναι και οι συνομιλητές μας, είναι οι επαφές μας τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να ε, συζητήσουμε ε, τις βελτιώσεις που μπορούμε να κάνουμε στις εκθέσεις τις οποίες υποβάλλουμε και προωθούμε. Σας είπα ότι η ζωή μας εξαρτάται από τη, τα σωστά συμπεράσματα, από τη σωστή, καλή ποιότητα των εκθέσεων που υποβάλλουμε, δηλαδή από την ποιότητα των φακέλων και το, την ολοκλήρωση των φακέλων. Ε, σκέφτομαι, έχω και την Ιταλία κατά νου, όπου μπορέσαμε πολύ νωρίς να συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές, να τους ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε, να τους στείλουμε τους φακέλους μας και να εξασφαλίσουμε την επιστροφή μεγάλων ε, ποσών χρημάτων, μεγάλων κονδυλίων ε, που είχαν ε, καταχραστεί και ήταν μια επιτυχημένη συνεργασία αυτή. Κάθε φορά λοιπόν που ξεκινάνε, ξεκινά ένας φάκελος φροντίζουμε για την πολύ γρήγορη προώθησή του και υποβολή του στις αρμόδιες εθνικές δικαστικές αρχές. Άρα στην εργασία μας είναι καλή και οι ε, αρχές ελέγχου, οι ελεγκτικοί φορείς χρησιμοποιούν πολλές φορές και με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις προφορίες ε, που δίνουμε εμείς για να προωθήσουν ένα φάκελο, μια υπόθεση δικαστική. Όσον αφορά τώρα τις, τους ε, συνεργάτες μας, έχουμε περιορισμούς ε, στην επιλογή, γιατί εμείς όταν δίνουμε ένα φάκελο δεν μπορούμε να διαλέξουμε ποιος θα είναι ο συνομιλητής μας, με ποιον θα συζητήσουμε το φάκελο, διότι δεν θέλουμε να ε, πιστεύει κάποιος ότι εγώ ποτέ ας πούμε το, το, όνομα το δικό μου δεν θα αναφερθεί ποτέ και δεν με χρησιμοποιείται ποτέ ε, στα δικαστικά πλαίσια, με αγνοείται. Ε, δεν διαλέγουμε εμείς λοιπόν με, με ποιους θα, θα μιλήσουμε, με ποιους θα έρθουμε σε επαφή, εξαρτάται από τις δικαστικές αρχές, ποιον θα επιλέξουν. Τώρα ο, η εφαρμογή του ελέγχου, εάν τον έλεγχο θα πρέπει να τον κάνουν οι αρχές που δαπανούν και τα χρήματα. Γιατί δεν είναι εμά βασικό ε, έργο να... Εμείς δεν καθορίζουμε ποιος θα δαπανίσει και θα δώσει τα χρήματα που. Εκ των υστέρων επεμβαίνουμε. Ε, βεβαίως ερχόμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους γενικούς ε, διευθυντές και τους ενημερώνουμε για τι έχει γίνει με τις πιστώσεις που διέθεσαν. Δεν τους ελέγχουμε βεβαίως εμείς. Ε, ελέγχουν, όπως σας είπα, οι, οι προϊστάμενες ελεγκτικές αρχές μου. Εάν σε μία υπόθεση, έχουμε μία εταιρεία, εμπλέκεται μία εταιρεία, μπορούμε να, να υποδείξουμε στις ελεγκτικές αρχές, κοιτάξτε, εδώ κάντε έναν έλεγχο στην εταιρεία αυτή, ερχόμαστε σε επαφή δηλαδή με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές ή με τις ε, διευθύνσεις της Κομισιόν και λέμε κάντε έναν έλεγχο τι γίνανε τα λεφτά αντιμετωπίζουμε καθημερινά ελεγκτικά προβλήματα διότι πρόκειται περί ευρωπαϊκών χρημάτων. Βεβαίω, τον πρώτο λόγο τον έχει η εθνική δικαιοσύνη και οι εθνικές αρχές δίωξης. Μπορούμε να βοηθήσουμε την παροχή πληροφοριών, τις εθνικές αυτές αρχές, οικονομικής φύσεως συνήθως πληροφορίες, Όπως σας είπα από την αρχή των, της παρέμβασής μας, βοηθούμε τις αρμόδιες αρχές να αυτοβοηθηθούν. Για την έκθεση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Παρακαλώ. Κύριε Μπρόνερ, συγγνώμη, σα ξαναδίνω το λόγο για την έκθεση τη Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Νόμιζα ότι πρέπει να απαντήσω και άλλη ερώτηση και δεν σας πρόσεχα. Συγγνώμη. Πρέπει τώρα να σας παρουσιάσω την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μου ζήτησε ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Κάλλας, να σας παρουσιάσω σήμερα την έκθεση αυτή την έκθεση του άρθρου 280 σε εσά, έτσι την αποκαλούμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι νεοφορμένοι να κατανοήσουν γιατί υπάρχουν δύο εκθέσεις και γιατί διαφέρουν μεταξύ των και γιατί αλλάζει, άλλαξα και γλώσσα, διότι είναι μια άλλη έκθεση και δεν είναι άμεσα δική μας ευθύνη. Είναι μια έκθεση την οποία η Όλαφ ετοίμασε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι διτός ο ρόλος μας εδώ. Το άρθρο 280 της συνθήκης λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συντονίζουν τις δράσεις τους προκειμένου να προστατεύσουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταπολεμήσουν την απάτη και τις άλλες ε, παρατυπίες που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό. Επομένως, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων είναι θέμα κοινή ευθύνη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχει πάντα κοινή ευθύνη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Συνεπώς, Βάσει αυτού του ίδιου άρθρου, κάθε χρόνο η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ετοιμάζουν από κοινού μία έκθεση για την προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η έκθεση αυτή παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που αφορούν υποθέσεις απάτης και άλλες παρατυπίες. Τα στατιστικά στοιχεία αυτά είναι, όπως ξέρετε, μεγάλο ενδιαφέροντος και για ε, εξωτερικούς παράγοντες, αλλά πρέπει να σας επιστήσω την προσοχή, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διότι οι εκθέσει παρατυπιών στι περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μια απλή παράληψη από πλευράς υπηρεσιών και να μην είναι απάτη που είναι ποινικά κολάσιμο δίκημα. Επίσης, η υποψία απάτης δεν είναι απαραίτητα απάτη και δεν επιβεβαιώνεται απαραίτητος από το δικαστήριο. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης τα νέα μέτρα που έχουν λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα, αλλά πρόκειται απλώς για παραδείγματα. Ε, αναφέρονται τα πάντα, διότι κάποια πράγματα ε, είναι απλά καθημερινή ρουτίνα και τα παρουσιάζουμε ε, μια φορά, δεν τα γράφουμε συνεχώς. Εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο κάθε χρόνο υιοθετεί ψήφισμα για την καταπολέμηση της απάτης ε, και το ίδιο κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Όλαφ. Ενώ το Συμβούλιο δείχνει πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον. Φαίνεται λοιπόν ότι ε, αυτό είναι ένα θέμα που εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για αυτή την προσέγγιση γιατί υποστηρίζει τα μέτρα μας. Στην έκθεση του άρθρου 280 που σας παρουσιάζω σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μια θετική συνέχεια στο αίτημα που ε, εξέφερσαν στην ε, έκθεση Μουζότο του 2008 και παρουσίαζε μια εικόνα των ε, εξουσιών και της οργάνωσης των αρχών των κρατών μελών που αφορούν σε θέματα καταπολέμησης απάτης και το συντονισμό τους με την Όλαφ, καθώς επίσης και μια εκτεταμένη ανάλυση της, των κανόνων πειθαρχία ε, που ε, χρησιμοποιούνται ε, για τις παρατυπίες στα κράτη-μέλη. Επισημαίνεται ότι βελτιώνονται ουσιαστικά τα συστήματα των κρατών μελών, κυρίως λόγω της μηχανογράφησης των συστημάτων και θα έχουμε και την εισαγωγή ενός συστήματος αναφοράς παρατυπιών μέσω διαδικτύου του IMS. Και Βέβαια χρειαζόμαστε περισσότερη ε, βοήθεια, χρειαζόμαστε και τη δική σας υποστήριξη, ώστε όλα, όλες οι παρατυπίες ε, βάσει των κανόνων να παρουσιάζονται, διότι έτσι θα έχουμε την καλύτερη εικόνα. Ε, δεν μπορούν κάποια κράτη-μέλη απλά να λένε, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία είναι στην κορυφή. Ναι, είναι στην κορυφή γιατί είναι διατεθειμένοι να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να μας πούνε τι πάει στραβά. Τώρα, πέραν των συγκεκριμένων θεμάτων που μόλις σας ανέφερα, να σας δώσω και μια εικόνα των βασικών στατιστικών τάσεων που αφορούν την απάτη και τις παρατυπίες. Τα συνολικά στοιχεία για το 2008 καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των παρατυπιών αυξήθηκε για τα διαρθρωτικά ταμεία και για τα ταμεία συνοχής, για τα ταμεία προένταξης και τις άμεσες δαπάνες και μειώθηκε για τη γεωργία και τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους. Οι συνολικές ε, οικονομικές επιπτώσεις που εκτιμούνται για τις δαπάνες μειώθηκαν από το 1 24 εκατομμύρια το 2007 στα 783,2 ε, εκατομμύρια ευρώ το 2008. Μειώθηκε σε όλους τους τομείς με εξαίρεση τις άμεσες δαπάνες και τα προεταξιακά ταμεία. Για τα προεταξιδετικά ταμεία ο αριθμός των νέων περιπτώσεων και τα ποσά ε, τα οποία αναφέρθηκαν είναι τα υψηλότερα που έχουμε μέχρι τούδε. Ο αριθμός των περιπτώσεων αυξήθηκε κατά 58%. Είχαμε 523 περιπτώσεις το 2008 η αύξηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα και ενισχυμένων ελέγχων στο τέλος του κύκλου των ε, ε, προγραμμάτων, του αυξαμένου αριθμού των χωρών που συμμετέχουν και ε, της μεγάλης ποικιλομορφίας προενταξιακών προγραμμάτων βοήθειας που εφαρμόζονται οι οικονομικές επιπτώσεις για τους παραδοσιακούς ήρους πόρους ε, μειώθηκε από τα 401 εκατομμύρια ευρώ το 2007 στα 351 εκατομμύρια ευρώ το 2008. Το συνολικό εκτιμόμενο, να επισημάνω, υπογραμμίσω εδώ το εκτιμόμενο ε, οικονομικές επιπτώσεις των περιπτώσεων όπου έχουμε υποψίες απάτης, μειώθηκαν και για τις δαπάνες ε, και για τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους. Τέλος, θα ήθελα να σας πω λίγα πιάγματα που αφορούν στα κύρια μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Να πω και κάτι για την πρόταση 2000 για το 1073 να αναφέρω και την ε, συμφωνία του Λίχτενστάιν, η οποία δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά θα καθορίσει προδιαγραφές για τις μελλοντικέ συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως το Μονακό και κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο Κοφίν ε, θα βάλει μια τελεία στο όλο θέμα, διότι πρέπει πλέον να γίνει. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για μένα είναι ότι ζήτησαν όλο και περισσότερα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον τη συμφωνία και λένε «Ω Χριστέ μου, μπορούμε να το υπογράψουμε αυτό». Πλέον είναι πάρα πολλά αυτά που μας ζητάτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η κατάσταση. Για μήνες ολόκληρους μας ζητούσαν περισσότερα και αυτή τη στιγμή του σοκάρει αυτό που μας ζήτησαν. Το Λίχτενστάιν ε, έχει συμφωνήσει και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση. Ελπίζω να βρουν μια λύση εντός του μηνός Οκτωβρίου για αυτή την ε, κατάσταση που δημιουργήθηκε. Είχαμε επίσης και κάποια μέτρα προκειμένου να προστατεύσουμε το νόμισμά μας, κυρίως ε, την παραποίηση, τα μεταλλικά νομίσματα. Είναι θέματα τα οποία είναι πολύ ε, γνωστά, υπάρχουν και στις ιστοσελίδες. Θέλουμε να προστατεύσουμε χαρτονομίσματα και μεταλλικά νομίσματα και άλλες ε, παρατυπίες. Αυτά λοιπόν, εν συντομία, ε, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση σε όλες τις γλώσσες είναι αρκετά σύντομη. Υπάρχει μια σύνοψη και να σας πω ότι κυρίως ε, για τον εισηγητή υπάρχουν δύο παραρτήματα τα οποία διατίθενται μόνο στα αγγλικά και αφορούν αποκλειστικά και μόνο στατιστικά στοιχεία για να τα επεξεργαστείτε. Έτσι έχει η κατάσταση. Δεν μπορούμε δυστυχώς να μεταφράσουμε όλη την έκθεση. Α, συγγνώμη, μόλι μου είπαν ότι τα παραρτήματα θα είναι σε τρει γλώσσε, αλλά και πάλι οι περισσότεροι από εσά δεν θα είστε ικανοποιημένοι γιατί δεν έχουμε όλε τι γλώσσε και έχουμε μόνο τρει. Έτσι έχει κατάσταση όμω. δεν έχουμε τη δυνατότητα να μεταφράσουμε το σύνολο τη έκθεση ε, συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων, διότι είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, αλλά ε, ελπίζουμε να σας βοηθήσουν οι τρεις αυτές γλώσσες. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος βουλευτής που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Παρακαλώ. ich, äh, bin auch Εγώ είμαι νέος. Πρέχομαι από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρέπει να συνηθίσω. Να συνηθίσω τα δεδομένα εδώ, Δηλαδή, ότι η υπηρεσία καταπολέμησης απάτης υποβάλλει ε, μια έκθεση στην Κομισιόν. Είναι δομές με τις οποίες δεν έχω εξοικειωθεί ακόμα. Α, φαντάζομαι ότι το σύστημα είναι δοκιμασμένο και λειτουργεί. Η απάτη είναι μια, ένα εσωτερικό ζήτημα και εξαρτάται, ε, βασίζεται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία καταπολέμησης της ε, απάτης και ενίσχυσης διαφάνειας έχουμε ε, στο ίντερνετ ε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε ε, όλες τις δραστηριότητες της περιφερειακής, της γεωργίας, του γεωργικού τομέα, αλλά στα διαφορετικά ταμεία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε και η δημοσιοποίηση των, πιστώσεων για τα διαφορετικά ταμεία είναι πάρα πολύ ελλειπή. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Ορισμένα στοιχεία που δημοσιεύονται αναφέρονται σε συγκεκριμένε περιοχές, αλλά δεν βοηθούν ε, τα συμπεράσματα που θέλουμε εμείς να συνάγουμε για τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται. Χρειάζεται λοιπόν να καλύψουμε αυτή, αυτά τα ελλείμματα, διότι ε, ε, πρέπει να επιβάλλουμε μία διαφάνεια στις διαφορετικές πιστώσεις, ώστε να αποφύγουμε Φεύγονται και να προλαμβάνονται οι μεγάλες απάτες που γίνονται σε αυτό το τομέα. Επίσης, ε, οι στόχοι, πρέπει να έχουμε διαφάνεια και στους στόχους που θέτουμε για την περιφερειακή πολιτική. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς τα διαστροτικά ταμεία θα εφαρμοστεί η πρωτοβουλία αυτή ε, της διαφάνειας. Ο κύριος Μπρίνερ οι δομές της Ευρώπης είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Αλλά δεν βλέπω ε, κανένα πρόβλημα με την υποβολή μιας εκθέματος ε, του Αντιπροέδρου της Κομισιόν. Εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας τα οποία μας ζητούνται και βάσει τις ε, συνθήκες και της συνθήκης, η Κομισιόν μαζί με τα κράτη-μέλη συντάσσει την τελική έκθεση. Άρα λοιπόν η δική μας έκθεση είναι υποβοηθητική και παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που χρειάζεται η Κομισιόν για να τσεκάρει ε, για να κάνει μια γενική επισκόπηση και καταγραφή της κατάστασης και να παρουσιάσει τα συνολικά στοιχεία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μέχρι τώρα Πολλές φορές έχουν υπάρξει επικαλύψεις ε, εργασίας, δεν μας έχουν ε, ενοχλήσει ή ιδιαίτερα στεναχωρήσει. Ε, είναι σαν να κάνουμε ένα διπλό έλεγχο αν θέλετε και μάλλον θετική είναι αυτή, η, αυτό το γεγονός. Η ουσία είναι ότι προσπαθούμε να ενσωματώσουμε, να βοηθήσουμε στην ενσωμάτωση και των δικών μας ε, στοιχείων. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τη διαφάνεια των διαθροτικών πιστώσεων. Ίσως μπορούν οι συνάδελφοι της Κομισιόν να βοηθήσουν αν θέλουν. Ε, θα απαντήσω γραπτός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω με συγκεκριμένα στοιχεία για τη διαφάνεια ε, στον έλεγχο των διαθροτικών πιστώσεων. είναι ένα, ένα, πλαίσιο το οποίο καλύπτει την Κομισιόν. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή εγώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή για το σύνολο των τοποθετήσεών του. Θα ήθελα να συμφωνήσω με κάποιους από τους προλαλήσαντες συναδέλφους μου για το θέμα της ανεξαρτησίας σας. Το γεγονός ότι μιλάτε εν ονόματι της Κομισιόν είναι ένα τεκμήριο μη ανεξαρτησίας. Μια και σημαίνει ότι α, είσαστε υποταγμένοι στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα παρουσίαζε είτε η ίδια είτε μέσω ενός προσώπου της ε, την έκθεσή τη. Την έκθεση της Κομισιόν, την οποία παρουσιάσατε εσείς. Αυτό το λέω εν είδη εισαγωγή. Δεν θέλω να αμφισβητήσω ακριβώ την εξαρτησία σα, αλλά νομίζω ότι μπροστά σε ένα πολιτικό όργανο όπω το δικό μα, γιατί το δικό μα καθήκον τη Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού είναι να ελέγξουμε την εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία είναι η Κομισιόν, η οποία θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί μα. Έτσι, είναι παρένθεση, την κλείνω. Επίση, θλίβομαι για το γεγονό το εξή. Είναι κρίμα που σε αυτή την έκθεση που όπως είπατε και εσείς κύριε Γενική Διευθυντά, μιλάει για το άρθρο 280 προστασία των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Είναι κρίμα λοιπόν που η Κομισιόν προσθέτει στην, στον τίτλο της έκθεσης καταπολέμηση της απάτης. Είναι κρίμα γιατί δίνουμε έμφαση στην καταπολέμηση της απάτης ενώ αυτή η έκθεση έχει μία πολύ πιο ευρία λογική. Και η διοίκηση που διευθύνεται είναι αυτή που καταπολεμά την απάτη, γιατί ονομάζεται Οργανισμός Καταπολέμησης της Απάτης. Δεν μ' αρέσει λοιπόν ο τίτλο τη έκθεσης. Να εκφράσω και μια άλλη δυσαρέσκεια που την είχα εκφράσει και στην απαλλαγή του περασμένου έτους. Ε, δηλαδή, σε όλες αυτές τις ε, υποθέσεις μάλλον μπερδεύουμε τις απάτες, τις παρατυπίες και όλο και περισσότερο προσθέτουμε και τις υπόνοιες απάτης. Και μια μέρα θα προσθέσουμε και τι υπόνοιε παρατυπία. Εμεί οι βουλευτέ, ξέρουμε γιατί υπάρχουν παρατυπίε. Έχουμε κανονισμού που είναι πάρα πολύ περίπλοκοι. Και επειδή είναι πάρα πολύ περίπλοκοι, τα κράτη-μέλη ή οι δικαιούχοι οι τελικοί κάνουν λάθη. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό να καταπολεμήσουμε την απάτη από το να διαπιστώσουμε μία πλειάδα παρατυπιών, όπως το κάνει πάρα πολύ καλά το ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα να διακρίνουμε μεταξύ παρατυπιών και η εμπειρία είναι το σύνολο το, της πείρας. Δεν είναι λάθος να κάνουμε, δεν είναι ασύνηθες μάλλον να κάνουμε λάθη. Υπάρχει βέβαια η απάτη κάτι που είναι πολύ σοβαρό γιατί υπάρχει το στοιχείο της πρόθεσης. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σε αυτή την έκθεση μιλάτε για την προστασία των οικονομικών συμφερόνων και την καταπολέμηση της απάτης. Για το 2008 μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο αριθμός των απατών τι πραγματικέ απάτε, όχι τι υπόνοιε. έτσι, τον αριθμό των απατών και το ποσό που αφορούν αυτέ οι απάτε. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ähm, να επαναλάβω. Είναι. Όλαφ έχει, όπως σας είπα, γενικά μία θετική ε, αξιολόγηση των εργασιών της και γι' αυτό δουλεύουμε και για την Κομισιόν και η φωνή της Όλαφ είναι ο διευθυντής της. Ε, Γι' αυτό ακριβώς υποβάλλουμε και αυτή την έκθεσή μα στην Κομισιόν. Εμείς έχουμε όλες τις πληροφορίες, όλα τα στοιχεία. Είμαστε το κεντρικό σημείο, η καρδιά δηλαδή ε, της ενημέρωσης ε, όλων αυτών των στοιχείων που χρειάζονται στη Γενική Διεύθυνση, στο Γενικό Διευθυντή δηλαδή, για να έχει μια γενική εικόνα της κατάστασης. Και γι' αυτό όταν ο κύριος Κάλλας ο Αντιπρόεδρος με παρακαλεί να παρουσιάσω την έκθεση. Δεν αισθάνομαι ούτε ότι χάνω την αντικειμενικότητά μου, ούτε ότι θίγεται η αντικειμενικότητά μου, ούτε η τιμή μου που συνέταξε αυτή την έκθεση. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε αντικειμενικότητος, ούτε τίποτα άλλο με την υποβολή αυτής της έκθεσης ε, στην ε, Επιτροπή. Πολλές φορές έχω μιλήσει και εξ ονόματος ε, της Κομισιόν. Τώρα γιατί έχω αυτό τον τίτλο στην έκθεσή μου μπορώ να σας το εξηγήσω. Τα κράτη-μέλη θα ήταν ενθουσιασμένα να διαγράψουν το Fight Against Fraud κατά πολέμηση της απάτης. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα πολλές φορές. Α, όμως, ε, εκ παραδόσεως, αυτό το αντικείμενο της εκθέσεως είχε προβλεφτεί. Δηλαδή, από την πρώτη έκθεση μέχρι αυτή, γιατί δεν είναι η πρώτη έκθεση αυτή, έχουν ε, ε, προηγηθεί πολλές. Είχε αυτό τον τίτλο, αυτή την ορολογία. Η γερμανική μετάφραση της Όλαφ λέει «Η υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης» στα γερμανικά λέει Amt, υπηρεσία και η μια υπηρεσία στο, στη Γερμανία δεν επιτρέπεται να διεξάγει ποινικέ έρευνε με ποινικό περιεχόμενο που καταλήγουν δηλαδή στη, στο ποινικό δίκαιο. Διότι για, το ποινικό, για, για τις ποινικέ υποθέσεις είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη. Βλέπετε λοιπόν ότι δημιουργούνται τέτοια θέματα ορολογίας αν τα αναλύσουμε κυριολεκτικά. Είναι εκ παραδόσεως που έχουμε αυτό τον τίτλο. Εγώ αυτόν βρήκα όταν ανέλαβα το αξίωμά μου και αυτόν αναγράφω. Έτσι ήθιστε λοιπόν να κάνουμε. Διότι πάρα πολλές παρατυπίες οδηγούν σε απάτη όσον αφορά αυτά τα οποία είπατε, γενικά, ε, για τις ε, μεθόδους υποβολής εκθέσεων. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι. Υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα που θεωρεί τα πάντα ως παρατυπίες. Τα ονομάζει παρατυπίες και αν συνεχεία μετά από 10 ή 15 χρόνια όταν επιτέλους βγει απόφαση του, του δικαστηρίου το μετονομάζει σε παρανομία. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Γερμανία όταν επέμβουν οι οικονομικές υπηρεσίες ή η αστυνομία απευθείας ο φάκελος ονομάζεται ως ε, απάτη. απάτη. Ξεκινά λοιπόν στην Ελλάδα από παρατυπία και γίνεται απάτη, ενώ στην Ιταλία και στη Γερμανία απευθείας χαρακτηρίζεται ως απάτη. Ε, είναι θέμα σαφήνειας ε, της ορολογίας. Υπάρχει αυτή η σύγχυση, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτό. Ε, γι' αυτό σας είπα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν, στα στοιχεία, στα μεγέθη ας πούμε, τόσες υποθέσεις τέτοιου μεγέθους. Ε, δεν έχουμε βρει μια μέθοδο ε, απολύτως αντιπροσωπευτική. Σας είπα, υπάρχουν και παραδόσεις στα εθνικά πλαίσια. Μόνο όταν υπάρχει καταδίκη πλέον και κατηγορητήριο σαφές μπορεί να χαρακτηριστεί μια υπόθεση ως απάτη, ενώ μέχρι τότε ε, ορίζεται ως παρατυπία ή ατασταλία και έτσι δημιουργούνται στατιστικά προβλήματα. Ξαφνικά μία παρατυπία του 90, της δεκαετίας του 90, αλλάζει, μεταβάλλεται σε απάτη του 2000. Ε, τι γίνεται λοιπόν, η ίδια είναι, αλλαγή ονόματος, ορολογίας. Πρέπει να, πω, σας πω και στον Νικάλε, το συνάδελφός μου, ο οποίος είναι ενήμερος αυτής της συζήτησης, Κάποια στιγμή πρέπει να λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό της ορολογίας και του, της ονομασίας, αν θέλετε, του χαρακτηρισμού των υποθέσεων. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και ελπίζω να μην πλέξουμε τα αυγά και τα πασχάλια, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρούινερ και να πάμε στο σημείο 8 της Μέσης διάταξης. Δύο παρατηρήσεις. Οι διεθνοί κανόνες ελέγχου επί τους οποίους βασίζεται το ελεγκτικό συνέδριο και εσείς, και ο εσωτερικός σας έλεγχο καθορίζουν τι είναι λάθος και τι είναι απάτη. Οι, απατη... οι είναι λάθη. Εγώ έδωσα ένα ερώτημα. Δεν μου δώσατε απάντηση. Ποιος είναι ο αριθμό των απατών και το ποσό των απατών. Ίσως να μην έχετε απάντηση, αλλά πάντως δεν μου δώσατε μέχρι στιγμής. Aufgrund der statistischen Probleme möchte ich sie nicht gleich beantworten, sondern nochmal das genau. Δεν μπορώ να σας απαντήσω άμεσα. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ γραπτός επί τη βάση των στατιστικών στοιχείων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία, αλλά επειδή είσαστε πολύ σαφεί, θέλετε τι απάτη τις απάτες τον αριθμό των πραγματικών απατών, θα σα απαντήσω γραπτό και θα σα στείλω τα στοιχεία. Ευχαριστούμε. Σημείο 8 στην Αίσια Διάταξη, παρουσίαση της μελέτης κώδικας διοντολογίας των επιτρόπων για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Η κυρία Κρέσλε. Της δίνω το λόγο. Er? Ο κ. Μπλόμαϊερ. Εδώ είναι. Ωραία. Τώρα πώς προέκυψε αυτή η μελέτη. Διαπιστώσαμε καταρχάς ότι υπάρχουν κενά στον κώδικα δεοντολογίας ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν καλύπτονται διόλου και το επιβεβαιώνει αυτό η μελέτη. Ξέρω ότι είμαστε υποχρονική πίεση, αλλά το θέμα αυτό είναι λίγα σημαντικό, διότι για μας, για την ακρόαση των ε, ε, επιτρόπων, θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτός ο κώδικας διοντολογίας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μπλόμπερκ. Πρέπει υποχρεωτικά, είμαστε υποχρεωμένοι να διευρύνουμε τον κώδικα και να τον ενημερώσουμε, να τον επικαιροποιήσουμε. Πρέπει να πούμε ότι διάφορα ταξίδια, διάφορα δώρα που δίδονται, είναι δώρα, είναι, δεν είναι, είναι σωστά, δεν πρέπει να δίνονται, να τα δέχονται. Δεν υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για ορισμένε διαδικασίες. Γι' αυτό ο κώδικας ε, δεοντολογίας πρέπει να αναθεωρηθεί. Πρέπει να αναθεωρηθεί. Καταρχάς πρέπει να ορίσουμε εκ νέου τι είναι δώρο, τι θεωρείται ως δώρο και όχι υλικό ή άϊλο δώρο, ας πούμε μία κορνίζα ή ένα ταξίδι. Επίσης, ε, πότε υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης, ποιος χαρίζει τι σε ποιον πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τι στοιχεία πρέπει να δηλώνονται, τι πρέπει να δηλώνουν οι επίτροποι, όταν λέμε οικονομικά συμφέροντα, financial interest, κάθε επίτροπος ερμηνεύει ε, τη δική του ερμηνεία τον όρο αυτό, την ορολογία αυτή. Να έχουμε λοιπόν ενιαίους ορισμούς. Και τι εννοούμε με συμφέροντα. Υπάρχει αντίφαση συμφερόντων εδώ. Υπάρχουν δραστηριότητε ενέργειες που είναι κατά των συμφερόντων. Ποια είναι τα ιδιαίτερα συμφέροντα τα οποία πολλές φορές εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα που λέμε οι επίτροποι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επακριβείς ορισμούς για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τον κώδικα διοντολογίας. Γι' αυτό ε, είμαι πολύ, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη που έχουμε τόσο λίγο καιρό. Πρέπει οπωσδήποτε να ρωτήσουμε την Κομισιόν και τη Γενική Γραμματεία πότε θα έχουμε μία εμπεριστατωμένη απάντηση για το πώς θα συνεχίσουμε με τον παλιό κώδικα δεντολογίας. Ο Μπαρόζο είπε ότι θα γίνει αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας αν έχει την, την, την ε, υποστήριξη όλων των υποτρόπων. Αλλά ε, το βρίσκω αυτό πολύ παράξενο, διότι η Κομισιόν είναι η υπεύθυνη για την, ε, ε, τον έλεγχο. και για τη σύνταξη ελαχίστων κανόνων. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Η Κομισιόν πρέπει οπωσδήποτε να μας απαντήσει. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπρούμερ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Παρακαλώ. Thank you very for the um, introduction. Um, the... Ευχαριστώ πολύ. Επειδή έχει προχωρήσει η ώρα, θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο γρήγορα γίνεται, παρουσιάζοντας τα κύρια σημεία που αφορούν σε αυτή τη μελέτη. Μια μελέτη που έγινε τους πρώτους πέντε μήνες του 2009 και μαζί με το Κέντρο Στατηγικής και Μελέτης Αξιολογήσεων ε, δώσαμε έμφαση στην εμπιστοσύνη ε, για τους στόχους και τη μέθοδο πολύ σύντομα και μετά θα φτάσω στα συμπεράσματα και στα, στις συστάσεις. Ε, ο σκοπός μας είναι να κάνουμε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του κώδικα διοντολογίας για τα μέλη της Κομισιόν, όπως ε, υιοθετήθηκε το 2004 από την Επιτροπή Μπαρόζο. Και από την αρχή ξεκαθαρίστηκε, μας ξεκαθαρίστηκε ότι αυτή η δουλειά θα έχει προστιθέμενη αξία μόνο εάν συνοδεύεται από πρακτικές συστάσεις. Κάναμε κάποια πρακτικά ερωτήματα, ε, κοιτάζοντας όλες τις ε, πλευρές του κώδικα, αν προωθεί την ε, διοντολογία αποτελεσματικά, αν προωθεί αποτελεσματικά την εμπιστοσύνη του κοινού, την αποτελεσματικότητα, αν δαπανώνται σωστά οι πόνοι. Κάναμε και ορισμένες μελέτες περιπτώσεων, κοιτώντα κυρίως το πλαίσιο της διοντολογία, σε ορισμένα από τα κράτη-μέλη, στη Δανία, στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και κοιτώντας την διεθνή εμπειρία που έχουμε στην ε, Παγκόσμια Τράπεζα και στο UNDP. Ε, ήρθαμε σε επαφή με, την, ε, με το Γενικό Γραμματέα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης, ο διαμεσολαβητής μας έδωσε κάποια στοιχεία. Συζητήσαμε τον ΩΣΑ για να καταλάβουμε καλύτερα τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ό,τι αφορά τη διοντολογία και την διαφάνεια διεθνώ, ε, Ήρθαμε σε επαφή ε, με κάποια πανεπιστήμια στη Σουηδία και στην Ελβετία. Έπειτα κάναμε λεπτομέρειες ερωτήσεις για τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο κώδικας διοντολογίας, δηλαδή την δήλωση συμφερόντο... την κοινοποίηση πολιτικών δραστηριοτήτων στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις ε, διατυπώσεις ό,τι αφορά την απασχόληση ε, πέρα από την, ε, τα, τις αρμοδιότητες στην Κομισιόν, ε, τα δώρα και κάποια οριζόντια θέματα, πώς εφαρμόζεται ο κώδικας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και, και στο εξωτερικό. Και κοιτάξαμε και το θέμα των κυρώσεων βεβαίως. Συνολικά θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα από αυτά που λέει ο κώδικας ε, διοντολογίας. Και μια και ο κώδικας ε, διατυπώθηκε αρχικά το 1999 επί Επιτροπής Πρόντι, στην πράξη έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. έχουν δοθεί πολλές κατευθυντήριες γραμμές, ε, πολλές πρακτικές έχουν δρεωθεί. Παρ' όλα αυτά, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πολλά, ότι πολλά ακόμα μπορούν να, βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, να εμποδίσουμε την σύγκρουση συμφερόντων, ε, την πρόθεση της ε, αξιοπρεπούς συμπεριφοράς, καθώς και της εμπιστοσύνης ε, του κοινού προς τα θεσμικά όργανα. Αυτό όμως επισύρει κάποιο κόστος. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τεράστια γραφειοκρατία για να παρακολουθούμε το θέμα της διοντολογίας. Πιστεύουμε ότι με τις συστάσεις που κάνουμε ε, μπορούμε να τις εφαρμόσουμε χωρίς ε, σημαντικό επιπρόσθετο κόστος. Τελικά φτάσαμε σε 28 συστάσεις και στο παράρτημα της μελέτης μας αναφέρουμε σαν κατάλογο ε, σύντομα και με μια σύντομη εξήγηση τις συστάσεις αυτές. Αφορούν κυρίως τη συμπλήρωση των διατάξεων του σημερινού κώδικα και την επισημοποίηση κάποιων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί εκτός του κώδικα, ε, από τις οποίες θα μπορούσε να υποφεληθεί ο κώδικας, αν τις ενσωμάτωνε. Επίσης, τώρα που ο κώδικας ε, έχει συσσωρεύσει κάποια χρόνια πίσω του, ε, υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Αναθεωρήθηκε βέβαια από την Επίτροπη του Μπαρόζο το 2004, αλλά στο μεταξύ ε, σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει πάρα πολλά. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές που έχουν αλλάξει και μπορεί να υποφεληθεί από αυτές ο κώδικας. Και εκεί που πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά, είναι το τελευταίο, είναι ότι θα έπρεπε να δημιουργηθούν κάποιες δομές ε, εφαρμογής ε, των όσων λέει κώδικας. Τώρα, για τις συστάσεις. Στη δήλωση συμφερόντων. Είναι από τα βασικά εργαλεία του κώδικα διοντολογίας. Ίσως ε, δηλώνουμε δηλαδή τις εξωτερικές δραστηριότητες, δηλώνουμε τα οικονομικά συμφέροντα, οι επίτροποι δηλαδή. Αυτό είναι χρήσιμο εργαλείο, μόνο όμως αν εξασφαλίζει ότι, πρέπει ότι είναι κατανοητή η, η οδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναγνώσκοντας τον κώδικα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναφέρονται και οι στόχοι των οργανισμών στους οποίους ενδεχομένως δουλεύουν οι επίτροποι. Υπάρχουν μια σειρά από επιτρόπους που το κάνουν αυτό και νομίζουμε ότι δίνουν ένα καλό παράδειγμα γιατί πραγματικά ε, έτσι υπάρχει σαφήνεια στον κώδικα. Επίσης συστήνουμε όλα τα οικονομικά συμφέροντα να αναφέρονται, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, αν θέλετε, και του παθητικού. Είναι διεθνής πρακτική αυτή σήμερα. Βεβαίως, είναι, υπάρχει και ένα κατόφλι πάνω από το οποίο δηλώνουμε τα, τα οικονομικά μας συμφέροντα, όχι τα ίσονο σημασία οικονομικά συμφέροντα. Επίσης και εδώ υπάρχει η διεθνής πρακτική ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να επικαιροποιούνται όχι μόνο όταν αλλάζει κάτι, αλλά σε αιτήσια βάση. Σε ό,τι αφορά το ποιο δηλώνει τι, ε, πιστεύουμε ότι όπως και οι σύζυγοι θα πρέπει και τα ανεξάρτητα παιδιά αλλά και οι σύντροφοι να δηλώνουν και αυτοί τις σχετικές πληροφορίες. Και επίσης ε, συστήνουμε να εισαχθεί μια ηλεκτρονική μορφή δήλωση των συμφερόντων. Σε ό,τι αφορά την πολιτική δραστηριότητα, ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο στοιχείο του κώδικα. Η πεποίθησή μας είναι ότι η ανεξαρτησία που, που απαιτεί η συνθήκη από εθνικά συμφέροντα μπορεί να, εγγυηθεί, να την εγγυηθούμε αποτελεσματικά αν περιοριστούμε ε, σε μια παθητική συμμετοχή, ας πούμε, σε κάποιο πολιτικό κόμμα σε εθνικό επίπεδο. Μια άλλη δυνατότητα βελτίωσης του κώδικα σε ό,τι αφορά την πολιτική δραστηριότητα είναι να υπάρχει μεγαλύτερη σαφάνεια σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για να αποφασίσουμε η εξωτερική πολιτική δραστηριότητα είναι συμβατή με, τη, με το λειτουργήμα του Επιτρόπου, με το αξίωμα του Επιτρόπου και να δούμε τι σημαίνει διαθεσιμότητα ε, με έτσι επίσημους όρους. Ό,τι αφορά τη διαφάνεια, θα ήταν επωφελές αυτές οι αξιολογήσεις ε, να δημοσιοποιούνται. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και να έχουμε και κάποιες προθεσμίες για να δηλώνουν οι επίτροποι τις ε, πολιτικές δραστηριότητες. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση μετά την ε, λήξη της περίοδου, όπου το άτομο είναι επίτροπο, Θα πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση τη συμβατότητα τη όποια απασχόλησης. Ε, θα πρέπει να γίνεται αυτό και για λόγους διαφάνειας, όπως είπα και προηγουμένως. Επίσης θα πρέπει να δημοσιεύονται αυτέ οι αξιολογήσει, πάλι για λόγους διαφάνειας. Επίση έχει νόημα να επεκτείνουμε την ε, περίοδο περιορισμού μετά την πάυση Τη δραστηριότητα Επιτρόπου σε δύο χρόνια. Σε ό,τι αφορά το μητρό δώρων, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι δώρο και να συμπεριλάβουμε εδώ και τη φιλοξενία, τον όρο της φιλοξενίας στον ορισμό των δώρων. Επίσης, ε, καλό θα ήταν να υπάρχει μια πολιτική κανένα δώρο σε ό,τι αφορά δώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης η, καταγωγή, η προέλευση των δώρων που προέρχονται από πηγές εξω... εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναφέρεται. Ε, δεν έχει νόημα να έχεις μια... ένα μητρό δώρο αν δεν μπορείς να αξιολογήσεις τη σύγκρουση συμφερόντων γιατί δεν ξέρεις από πού προέρχεται το δώρο από την, Ευρωπαϊκή... από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα ταξίδια και το προσωπικό. Ε, πολλές ε, χώρες έχουν εμπειρία για τη δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών. Τα ταξίδια θα πρέπει να δημοσιεύονται ετησίω με λεπτομέρειες και νομίζω ότι καλό θα ήταν για τον κώδικα να έχει σαφείς συστάσεις ό,τι αφορά την αποχή από αποφάσεις που παίρνουν μέλη της οικογένειας. Ο Γενικός Γραμματέας έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ ε, και γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα του κώδικα διοντολογίας. Ήδη από την Επιτροπή πρώτη. υπήρχε μια ομάδα ε, συμβουλευτική για τα πρότυπα της δημόσιας ζωής. Υπάρχει και τώρα μια ad hoc Επιτροπή Διοντολογίας ε, η οποία θα μπορούσε να διευρυνθεί. Ο χειρισμός το, της σύγκρουσης των συμφερόντων. Σε ό,τι αφορά την Επίτροπο Κρούς, παραδείγματος χάρη. Ε, σε ό,τι αφορά την, το, τον κώδικα, συγγνώμη, την Επίτροπο Κρούς, νομίζω ότι θα πρέπει να διαδίδουμε ε, και να ενημερώνουμε κάπως ε, το πώς εφαρμόζεται ο κώδικας κάθε χρόνο και να υπάρχει μια ορατότητα ε, αυτού του κώδικα, μεγαλύτερη από ό,τι τώρα. Γιατί είναι δύσκολο να βρεθούν αυτές οι πληροφορίες. Και τέλος, παράπονα και κυρώσεις. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό μηχανισμοί, θα μπορούσαν να διευκρινιστούν αν υπάρχει μια αναφορά τον διαμεσολαβητή, α πούμε, στον κώδικα διοντολογία και σε μια αναφορά σε που προβλέπει η ίδια η συνθήκη. Και σε ό,τι αφορά τι μικρέ παραβάσει, παραδείγματο χάρη το, μην, το να μην ε, συμπληρώνει άλλε πληροφορίε κανεί ή το να μην τι ε, υποβάλει έγκαιρα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δημοσιοποιούμε τέτοιου τύπου παραβάσει για να είναι πιο αποτελεσματικό ο κώδικα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να είστε λίγο συνοπτικοί γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ο κύριος ε, Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ για τη σύντομη και Λίαν ε, πληροφοριακή σας παρουσίαση. Η Κομισιόν δεν είναι ο μόνος ε, φορέας αποφάσεων για, την, για τον κώδικα διοντολογίας και τις παρατυπίες ή παραβιάσεις του, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει εκδώσει αποφάσεις οι οποίες γίνονται σεβαστές από την μεγάλη πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών. Υπήρχε, μία περίπτωση ενός φαρμακείου όπου ο γαμπρός παντρεύτηκε την κόρη του φαρμακοποιού και του δόθηκε η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου. Λοιπόν... Nicht nur ε, πρέπει να ξέρουμε ότι σε, σε περιπτώσεις τέτοιες, ε, τέτοιων προτιμησιακών χειρισμών και παραβιάσεων είναι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αρμόδιο, όχι μόνο η Κομισιόν. Δεύτερο παράδειγμα που θέλω να αναφέρω είναι οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί έχετε αναφέρει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών οργανώσεων, όμως πρέπει να ασχοληθούμε έντονα με τις διασυνδέσεις μεταξύ ε, επιτρόπων και μη κυβερνητικών οργανισμών. Διότι αυτές ε, οι, αυτοί οι οργανισμοί πολλές φορές χρηματοδοτούνται μέχρι 80% από εμά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι κυβερνητικοί οργανισμοί ΜΚΟ, Οπότε υπάρχουν διάφορες, ε, διάφορα ευαίσθητα σημεία. Π.χ. η ανταλλαγή επιστολών. Τι γράφει ο, ο Επίτροπος στις ε, ΜΚΟ και τι απαντήσεις παίρνει. Ε, πρέπει να δημοσιοποιούνται οι επιστολές αυτές. Υπάρχει διαφάνεια. Σας παρακαλώ λοιπόν να υπάρξει ισότιμος χειρισμός των μη κυβερνητικών οργανισμών με αυτός των λόμπιστ, των εκπροσώπων των λόμπι. Η κυρία Ανδρέας. Thank you, Mr. Chairman. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Είναι πάρα πολύ σαφής και ακριβής όσον αφορά στις συστάσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί περίμενε τόσο καιρό για την αναθεώρηση αυτού του κώδικα διοντολογίας, διότι 10 χρόνια είναι πολύ καιρό. Επίσης, ένα από τα πιο ανησυχητικά συμπεράσματα που είδα στην έκθεσή σας είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν καλύπτεται από τον κώδικα διοντολογίας. Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό και ακόμα περισσότερο ανησυχητικό δεδομένου ότι μόλις επανεξελέξαμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα ήθελα και μια απάντηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Και η τρίτη ερώτησή μου, αυτήν δεν ξέρω σε ποιον να την απευθύνω, είναι τι γίνεται τώρα και πότε ακριβώς, πόσο σύντομα. Διότι ε, σύντομα θα γίνουν οι ακροάσεις όλων των επιτρόπων και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό ε, και πρέπει να το έχουμε αντιμετωπίσει στο μεταξύ. Ο κύριος Οντή. Πολύ σύντομα. Τα θεσμικά μας όργανα δεν προβλέπουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζει τον Α ή τον Β, Β Επίτροπο. Έχουμε ένα δικαίωμα ομαδικής μουμφής. Για το θέμα των κυρώσεων, που είναι βασικό σημείο, θα μπορούσαμε για βασικές, ε, βασικά προβλήματα να προβλέψουμε το Κοινοβούλιο να ξανακάνει την ακρόαση του Α ή του Β επιτρόπου, ούτω ώστε να εξηγηθεί ε, για ορισμένα πράγματα τα οποία διαπιστώσαμε, α πούμε, κατά τη διάρκεια τη άσκηση των καθηκόντων του. Ε, να εξηγηθεί σε κάποια σημεία τη συμπεριφορα του, α πούμε. Είχαμε και μια ερώτηση της κυρίας Σέν, η οποία απευθυνόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή είναι παρόν εδώ ο κύριος Λατσβέσκι. Εάν θέλετε να παρέμβετε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, President, and uh, for... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια που καταφέρετε να προφέρετε και το όνομά μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ω απάντηση λοιπόν στην κυρία Αντρέασαν, καταρχά γιατί περίμενε τόσο καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν περίμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα η Επιτροπή Μπαρόζο το 2004 αναθεώρησε τον κώδικα διοντολογίας και τον βελτίωσε. Όπως ε, γνωρίζουμε, πάντα υπάρχει χώρος για βελτιώσεις, ακόμα και στα βελτιωμένα κείμενα. Επομένως, ακόμα και στις κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κυρίου Μπαρόζο, αναφέρεται ότι έχει πρόθεση να αναθεωρήσει τον κώδικα διοντολογίας και θα το κάνει. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα γιατί θεωρήθηκε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν καλύπτεται από τον κώδικα διοντολογίας, καλύπτεται και πρέπει να τηρεί τους ίδιους κανόνες με τους υπόλοιπους επιτρόπους. Ωστόσο υπάρχει μία πτυχή στην έκθεση των συμβούλων που ακούσαμε η οποία απουσιάζει διότι η έκθεση ήταν για τον ίδιο τον κώδικα δεοντολογίας και είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή. Υπεράνω όλων είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην ξεχνάμε ότι οι επίτροποι είναι πολιτικοί και είναι υπόλογοι ενώπιον του Κοινοβουλίου. Επομένως, οι εξουσίες για τη διασφάλιση των δεοντολογικών κανόνων δεν είναι μόνο στα χέρια των επιτρόπων ε, μέσω του κώδικα δεοντολογίας, αλλά είναι και στα χέρια του Ευρωπαϊκού, Κοινοβουλίου ως νομοθέτη. Ελπίζω να σας κάλυψε η απάντησή μου. Πρέγω. Κύριε Γκρέσλα, ευχαριστώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν, επειδή είμαι εισηγήτρια. Θα, έχουμε, θα έχετε μία γνωμοδότηση πλήρη, όπου θα αναφέρονται οι απόψεις μας και οι συστάσεις μας για την αναθεώρηση του κώδικα διοντολογίας. Εφόσον μας το ζητήσετε θα το κάνουμε αυτό. Έχουμε τον επίσημο αλλά και τον άτυπο δρόμο που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Εγώ θα προτιμούσα την άτυπη οδό, αλλά αφού μας το ζητήσατε επισήμως, θα σας υποβάλουμε και επισήμως τη γνωμοδότησή μου. Δεν έχω παρατηθεί ακόμα από το, την άτυπη μέθοδο, αλλά για να την ακολουθήσουμε αυτή θα έπρεπε να υποχωρήσει η μία πλευρά. Θα σας παρακαλούσαμε να μας βοηθήσετε στο πώς θα θέλετε να διαμορφώσετε την εικόνα αυτού του κώδικα. Δεν έγινε αυτό μέχρι τώρα θα καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα λοιπόν στην Ολομέλεια και θα πρέπει οπωσδήποτε να κρίνουμε τι έγινε μέχρι τώρα και τι δεν έγινε. Εγώ θα ήθελα να αποφύγω αυτή την, να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας και να βγάλουμε τα άπλητά μας στη φόρα, να βγουν τα άπλητα στη φόρα γενικά, αλλά δεν το πέτυχα. Εφόσον δεν ακολουθήσαμε τον άτυπο δρόμο, θα πρέπει να περιμένετε την επίσημη γνωμοδότησή μας και το ψήφισμα. Σε κάθε προϋπολογισμό γίνονται τέτοιες συζητήσεις, σε κάθε απαλλαγή του προϋπολογισμού το ίδιο παιχνίδι παίζουμε. Αλλά δεν μ' αρέσει. Αυτή, αυτό το παιχνίδι που παίζεται κάθε φορά δεν μ' αρέσει. Δεν εξαρτάται από εμά. Να σας πούμε τι να κάνει το κοινοβούλιο. Όπως σας είπα, ο πρόεδρος υποσχέθηκε να αναθεωρήσει τον κώδικα συμπεριφορά διεντολογία. Και θα το κάνει. Είναι σαφές ότι η έκθεση των συμβούλων δεν αντιπροσωπεύει το 100% του, του, των αναγκών του νέου κώδικα. Δηλαδή δεν είναι ντε και σόνι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε για τη μεταρρύθμιση, ένα θεωριστού του κώδικα. Ε, κάνει μια ανασκόπηση της κατάστασης, κάνει ορισμένες συστάσεις, αλλά όπως και είπε και ο πρόεδρος, ε, πιστεύει ότι αυτός ο κώδικας θα αποτελέσει μια βάση αναφοράς που θα εμπνεύσει και άλλα θεσμικά όργανα. Όπως είπε και ο κ. Χατζημαρκάκης, θα πρέπει να μπορεί ο κώδικας διοντολογίας αυτός να εφαρμόζεται και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς. Δεν είναι λοιπόν η ευθύνη των συμβούλων να μας πούν τι θα γίνει, ούτε αυτοί θα αποφασίσουν. Πρέπει όμως να μελετήσουμε την εκθεσή τους, έτσι. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και όλο και περισσότερο αυξάνονται οι επιφυλάξεις μου πολλά χρόνια συμμετέχω στην, πολιτική, στην ευρωπαϊκή πολιτική και κατανοώ ότι το, το, το νομοθετικό έργο του σώματος αυτού τονίζεται, το τονίζει η Κομισιόν ή όταν δεν έχει σχέδια δικά της ή όταν δεν ξέρει πώς να προχωρήσει. Μετά από όλα αυτά που άκουσα πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση Έχω και ε, από το, την πολιτική μου ομάδα αρκετές εμπειρίες με τις ε, δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και στο παρελθόν ο πρόεδρος της Κομισιόν. Ε, υποστηρίζω την ε, πρόταση, αυτά που είπε τις παρατηρήσεις της κυρίας Αντρέασεν ότι ο ΜΕΝ πρόεδρος εκλέχθηκε, αλλά πολλές ακροάσεις που αφορούν επιτρόπους εκκρεμούν ακόμα. Οπότε τίθεται το ερώτημα, πρέπει στο, να δραστηριοποιηθούμε ε, στον κώδικα δεοντολογίας τώρα και τι, πώς θα τον εφαρμόσουμε εφόσον εκκρεμούν αυτές οι ακροάσεις τώρα βάσει ποιου κώδικα. Πάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, την παρουσίαση της μελέτης «Η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Γερμανία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο» Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπλομάιερ ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι δύο μελέτε που έγιναν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου, το ένα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, στη Γερμανία, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και η άλλη ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παρουσιάσω απευθεία τι συστάσει μα και για τι δύο, διότι έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ που δεν υπάρχει λόγο να τι διατρέξουμε μία προ μία τι παρουσιάσει. Okay. Ωραία, λοιπόν. Βάσει των όσων κάναμε σε αυτούς τους έξι μήνες, οι βασικές μας συστάσεις είναι να δώσουμε έμφαση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των δύο ταμείων, και του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο, σε έναν διάμεσο στάδιο και κυρίως να έχουμε ε, συγκρίσεις αναχώρα που είναι μία από τις αδυναμίες που διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί. Επίσης θα θέλαμε να προτείνουμε το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενισχύσει τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογηθεί το 2010, που είναι η χρονιά στην οποία θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα ε, βάσει αυτής της εργασίας. Είναι πολύ δύσκολο να το κρίνουμε, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε στη διάρκεια της μελέτης μας. Θεωρούμε το 2010 είναι μια καλή χρονιά να δούμε τι συνέβη, τι έχει βελτιωθεί. Έχουμε διαπιστώσει ήδη κάποιες βελτιώσεις. Ο κύριος ε, ε, Γκρένερ αναφέρθηκε σε κάποιες βελτιώσεις οι οποίες δεν απευθύνονται απευθεία στα διαρθρωτικά ταμεία. Στα διαρθρωτικά ταμεία είχαμε κάποιες βελτιώσεις ως προς τον όγκο των παρατυπιών ε, και έχει μειωθεί κατά 30% ο αριθμός των παρατυπιών. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο και θα πρέπει να δούμε και σε ποιο βαθμό ε, και ίσως και οι πιο αποδοτικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως διορθωτικά μέτρα, έχουν βοηθήσει τα αίτια ε, των παρατυπιών θα πρέπει να αναλυθούν εις βάθον. Ε, λέμε ότι έχουμε υψηλά ποσοστά παρατυπιών, δεν αναφέρεται τίποτα για την ποιότητα της ε, δημοσιονομικής διαχείρισης και του ελέγχου. Ίσως καλό θα ήταν να γίνουν αυτές οι συγκρίσεις και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μέσω δικτών για την ποιότητα και για την ένταση των ελέγχων που γίνονται στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα στις αιτήσει εκθέσεις, αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που εξετάσαμε στη μελέτη και φρονούμε ότι καλό θα ήταν να έχουμε περι, περαιτέρω καθοδήγηση στα κράτη-μέλη για την ε, συνολική ανάλυση των αποτελεσμάτων και εδώ ίσως θα μπορούσαμε, ε, δεδομένου ότι υπάρχουν πλέον περισσότερα κράτη-μέλη που δίνουν αυτά τα στοιχεία, να κάνουμε και μια κάποια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Τέλος, θεωρούμε ότι η Επιτροπή Επαφής που είναι ε, ο χώρος στον οποίο συναντούνται τα Εθνικά Ινστιτούτα Ελέγχου και οι Εθνικές Αρχές ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν να ενισχύσουν την συνεργασία τους, να δούμε πώς αναλύονται αυτές οι αιτήσεις εκθέσεις και η περαιτέρω ανάλυση των πληροφοριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για την ταχύτητά σας. Το τελευταίο σημείο, το οποίο εσείς θα μας το παρουσιάσετε. Κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με ενδιαφέρει το θέμα, γιατί το θέμα της αποτελεσματικότητας των ταμείων έχει πολλές ε, πτυχές και υπάρχουν και πολλές απόψεις. Γι' αυτό με ενδιαφέρουν, διότι από τέτοιες μελέτες ε, πολλές φορές ε, προκύπτουν αποτελέσματα που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ε, προβληματικά. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Μπλουμέγερ γιατί επιλέξατε περιόδους από το 2000 και μετά και δεν είδατε καθόλου το προηγούμενο χρονικό διάστημα, διότι εκεί είχαν περατωθεί οι έρευνες και ο κύριος Μπρούνερ μας παρουσίασε μία έκθεση του 2008 που περιέλαμβανε και στοιχεία από το 84 ε, μέχρι το 99. Γιατί λοιπόν δεν μελετήσετε ε, μία περίοδο που είναι κλειστή και μελετήσετε μία περίοδο που είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Θα είχαμε αποτελέσματα τα οποία θα ήταν πιο συνολικά διότι τα τρία κράτη-μέλη που ε, μελετήσατε, ούτως ή άλλως είναι παλιά κράτη-μέλη. Από το 84 μέχρι το 99 ε, λάμβαναν κονδύλια από τα ταμεία αυτά. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω γιατί στο παράρτημα 2 που έχετε τον κατάλογο των, ε, αυτών που χρησιμοποίησατε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, φαίνεται ότι ο αριθμός των ατόμων που έχετε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας ολόκληρος κατάλογος και ε, κράτη-μέλη που έχουν σημαντικές ε, εκτελέσεις προϋπολογισμού όπως είναι η Ισπανία και η Γερμανία φαίνεται να έχουμε μια διαβούλευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μόνο ελεγκτών. Δεν έχουμε τίποτα σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Υπάρχει θέμα εδώ αποτελεσματικότητας. Μου φαίνεται αντιφατικό για παράδειγμα να προκύπτει ως ε, σύνοψη να λέτε Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για την ε, υποστήριξη του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου Συνοχής. Δεν ξέρω αν οι πολίτες των χωρών αυτών, κυρίως οι πολίτες της χώρας μας, θα ε, ήταν ικανοποιημένοι με την αποδοτικότητα των δομών σε όλα τα σημεία, τις περιβαλλοντικές, τις θέσεις απασχόλησης που προέκυψαν. και υπάρχει και ένα συμπέρασμα το οποίο δεν είναι, λέτε ότι δεν είναι εναρμονισμένοι όλοι οι δείκτες. Εντάξει, αυτό είναι σαφέ, αλλά αν δεν είναι εναρμονισμένοι ω συμπέρασμα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να αποδείξουν ότι είναι περιορισμένη η αποδοτικότητα. Στην περίπτωση τη Γερμανία, για παράδειγμα, μιλάτε για 40.000 ε, επιχειρήσει ω στοιχείο αποτελεσματικότητα. Στην Ισπανία μιλάτε μόνο στο στόχο 2 για 2.000 θέσει απασχόληση και στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου Έχετε μόνο στόχο 2 και έχετε μόνο μία εκτίμηση η οποία μου φαίνεται ότι δεν ε, συνάδει με τα στοιχεία που έχετε για την Καταλωνία. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα, διότι οι συστάσεις και τα συμπεράσματα είναι ε, γενικά, γενικευμένα θα έλεγα και ε, υποτίθεται ότι έχετε κάνει μια μελέτη εις βάθος, όλα αυτά τα συμπεράσματα χρησιμοποιούνται ε, από αυτούς που θέλουν να είναι υπέρ, υπέρ των αποτελεσμάτων, αυτών που θέλουν να είναι κατά, κατά των αποτελεσμάτων και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι κυρίως ε, τα περιφερειακά ταμεία στις τρεις χώρες που μελετήσατε, ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι έχουν αποτελεσ... περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι πολίτες έχουν απορίες και έρχονται εδώ να επαληθεύσουν πώς λειτουργούν οι υποδομές μας δεν ξέρω λοιπόν ε, σε τι ανταποκρίνεται αυτή η περιορισμένη αποδυτικότητα σε εφαρμογή των ταμείων. Σε κάποια άλλα κρατημέλη μου φαίνεται ότι στη Γερμανία λειτουργούν πολύ καλά τα πράγματα και έχουν ε, δημιουργηθεί πολλές θέσεις απασχόλησης. Κάπου λοιπόν αντιφάσκουν τα στοιχεία. Α, όταν τα αναλύετε μας λέτε ότι έχουμε συνδεματική συνεισφορά και μετά στη σύνοψη, που είναι αυτή που θα διαβάσει και όλος ο κόσμος, ε, το απόσπασμα, έχετε ε, κάτι το οποίο αντιβαίνει με όλα σας τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ähm, έχετε δίκιο. Όσον αφορά στις ε, χώρες μέλη, η περιορισμένη αποδοτικότητα, εγώ ζω στην Καστήλια Λαμάντσα και ξέρω πολύ καλά τι εννοείται με αυτό που μας λέτε. Η περίοδος λοιπόν που αναλύσαμε, κυρίως ε, το διάστημα 2000-2006, αυτό ήταν αυτό το οποίο μας ανατέθηκε. Μας ζήτησαν να αναλύσουμε, να εξετάσουμε αποκλειστικά αυτό το χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες σε αυτή τη ε, μελέτη, το καταλαβαίνετε αυτό, καλύπτει πολλές χώρες και καλύπτει και πολλά ερωτήματα πολύ σημαντικές ερωτήσεις, οι οποίες ε, ίσως θα έπρεπε να είναι αντικείμενο μιας πιο εις βάθος μελέτης. Ε, το ξέρετε κι εσείς ε, τι πόρους διαθέτουμε στα πλαίσια αυτών των μελετών. Είναι πολύ περιορισμένοι οι πόροι μας. Όσον αφορά τώρα στην αποτελεσματικότητα, ίσως η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε να μην είναι η κατάλληλη. Αυτό που θέλαμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια κάποια έλλειψη δεδομένων ως προς την αποτελεσματικότητα, που μας επιτρέπουν να εξάγουμε συμπεράσματα κυρίως στα κράτη-μέλη τα οποία επιφολήθηκαν των ε, ταμείων σε αυτό το χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πολύ καλά ε, στοιχεία, για παράδειγμα στην Ισπανία για τις υποδομές που αναφέρθηκαν ε, σε άλλες χώρες σε θέματα καινοτομία, καινοτομίας, ποικίλουν τα αποτελέσματα. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που μας επιτρέπουν να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών και σίγουρα μεταξύ όλων των κρατών μελών ε, σε πολύ καλό, με πολύ καλό τρόπο συνολικό. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία, αλλά ε, επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει και κάποια απόπειρα σύγκριση. Οι μέθοδοι αξιολόγηση είναι τελείω διαφορετικοί μεταξύ των κρατών μελών. Οι δείκτε είναι πάρα πολύ ασθενεί και ξέρω ότι ε, η προσπάθεια αξιολόγησης ε, κατόπιν εορτής είναι εξελίξη. Εγώ εργάζομαι με πάρα πολλές τέτοιες ε, εξπόστ αναλύσεις οι οποίες δεν, θα, δεν νομίζω ότι θα δώσουν πολύ καλά στοιχεία γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Η απόδειξη λοιπόν της αποτελεσματικότητας, κυρίως μιας αποτελεσματικότητας που θα μας επιτρέψει να συγκρίνουμε μεταξύ κρατών μελών είναι περιορισμένη. Αναγνωρίζω ε, ότι ίσως ήταν λάθος η διατύπωση εδώ. Δεν ξέρω αν σα ε, κάλυψα. Ευχαριστώ. Ε, εκφράσατε ορισμένε ε, κρίσει για ένα παλιότερο διάστημα. Πιστεύω όμω ότι Καλά είπα ότι αν είχαμε και τη διαφάνεια στα τα ταμεία, στα διαθρωτικά όργανα, διαφάνεια επί των προγραμμάτων, τότε θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα τεράστιο βήμα πρόοδου. Δυστυχώς η εφαρμογή της ε, καινοτομίας ε, της πρωταβουλίας ε, διαφάνειας εφαρμόστηκε σε πολύ περιορισμένο εύρος ε, στον γεωργικό τομέα και σκεφτείτε με αυτή την, ε, την πρόθεση του θέματος της διαφάνειας τι πράγματα αποκαλύφθηκαν στον αγροτικό τομέα. Πολλά περισσότερα λοιπόν υποκρύπτονται στα, πίσω από το διαφορετικό πλαίσιο. είναι πάρα πολύ απαιτητικά τα διαφορετικά προγράμματα, πρέπει να καλύπτουν... Ε, Πάρα πολλά κριτήρια, καινοτομίε περί προστασία του περιβάλλοντος και πολλά άλλα στοιχεία. Εάν λοιπόν είχαμε ξεκινήσει από την περιφερειακή πολιτική και είχαμε πει ότι θα πάρετε τα χρήματα εάν μπορέσετε να μας αποδείξετε ότι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν ε, καλής ποιότητας νερό ε, ή ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση των δρόμων. Δεν θέσαμε όμως αυτά τα κριτήρια και γι' αυτό έχουμε δυσκολέψει τη ζωή μας. Και τέλος, κάθε φορά που κάτι πάει εντελώς τραβά σε ένα κράτος μέλος, τότε ξεκινάμε το μηχανισμό ε, αντιμετώπισης ε, της κρίσης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι νέους μηχανισμούς πρέπει να επιβάλλουμε, τι διορθώσεις και πρέπει να κάνουμε και κενά να καλύψουμε. Είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουμε με τα μούτρα κάθε φορά. Και τακτικά. Δεδομένου ότι συνεχώς ανακαλύπτουμε προβλήματα στη διάθεση και ε, στην απορρόφηση και στον τρόπο εφαρμογής των πιστώσεων που δίνουμε. Ενώ θα έπρεπε να είχαμε φροντίσει να εφαρμόζονται σωστά οι οδηγίες και οι κανονισμοί. Πιστεύω ότι έχουμε προχωρήσει, έχουμε τώρα νέους μηχανισμούς με τους οποίους μπορούμε να εφαρμόσουμε πολύ καλύτερα την οδηγία για τη διαφάνεια και όλο το πλαίσιο επιβολής των μέτρων διαφάνειας. Και με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Θέλω να σας θυμίσω γιατί έγινε αυτή η μελέτη. Έγινε αυτή η μελέτη, γιατί την αναθέσαμε, διότι στα έγγραφα εργασία της Κομισιόν από πέρσι έλεγε ότι αυτά τα κράτη-μέλη για τα οποία συζητάμε τώρα ε, είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να κάνουν αυτές τις παρατυπίες. Και γι' αυτό θέλουμε περισσότερα στοιχεία και ενημέρωση. Θέλαμε να ξέρουμε ποια και πού ακριβώς είναι τα προβλήματα στα κράτη-μέλη. Ευτυχώς σε λίγα κράτη-μέλη παρουσιάστηκε αυτή η διασύνδεση όταν υπάρχουν και σημειώνονται παρατυπίες πρέπει να ρυθμίσουμε και εμείς τις ε, ενέργειές μας. Πιστεύω ότι αυτή η μελέτη ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, τώρα όμως πρέπει να προχωρήσουμε την υπόθεση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν γνωρίζουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για την εφαρμογή των διορθωτικών προγραμμάτων στα κράτη-μέλη. Και αυτή η έλλειψη γνώσεων και εποπτείας πρέπει να μας απασχολήσει και στα επόμενα χρόνια. Ο κανονισμός λέει 2000-2006, προηγούμενος δηλαδή, και τα προβλήματα, πρέπει να κάνουμε μια γενική καταγραφή των προβλημάτων που σημειώθηκαν αυτό το διάστημα, αυτή την προηγούμενη εξαετία, για να κάνουμε τα πασίματα μασίματα. Εάν τώρα δεν πιστεύετε ότι αυτή η μέθοδος είναι σωστή, προτείνετε μας κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος μας, ότι πρέπει να πρώτα να κάνουμε καταγραφή και διαπίστωση και εν συνεχεία διόρθωση των προβλημάτων στο διαφορετικό τομέα και ταμεία. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ε, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε σε δύσκολη χρονική στιγμή, όπως συνέβη και πριν λίγους μήνες πριν. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα και συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την αποτελεσματικότητα, αυτή η συζήτηση είναι πολύ μακρόπνοη. Πώς θα τη μετρήσουμε, πώς θα μετρήσουμε την αποδοτικότητα της α β πολιτικής, ειδικά της πολιτικής συνοχής. Και εδώ μπαίνει το πρόβλημα των δικτών και της δυνατότητα να συγκρίνουμε ε, διαφορετικές μετρήσεις σε διαφορετικές χώρες. Μην ξεχνάτε ότι για κάθε πρόγραμμα έχουμε μία δέσμη δικτών που πρέπει να υπάρχει. Και όλα μας παραπέμπουν λοιπόν ε, στον α ή στο β δίκτυ του εκάστοτε προγράμματος. Αυτό είναι δύσκολο λοιπόν. Ε, Παραδείγματο χάρη, έτσι βλέπετε, μπορείτε να δείτε την επιρροή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, στο ΑΕΠ με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε για την αποδοτικότητα. Αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για την αποδοτικότητα ε, και πώς επηρεάζεται αυτή από λάθη ε, ή παρατυπίες. Είναι σωστό αυτό, κύριο Σοντή, ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτά για τα οποία μιλάμε. Τι θέλουμε, να αντιμετωπίσουμε την αποτελεσματικότητα με όρους ε, παρατυπίας, Γι' αυτό λοιπόν αυτή η μελέτη για μένα, και ίσω να κάνω λάθος, αφορά κυρίως την αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τις παρατυπίες και τις διορθώσεις τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα τμήμα τη συζήτηση όμως. Το άλλο τμήμα είναι η αποδοτικότητα σε ό,τι αφορά τις συνέπειες. Και αυτό το συζητούσαμε με την ε, Επιτροπή. Γιατί κάτι που μπορεί να είναι πολύ θετικό μπορεί να είναι γεμάτο από λάθη. Ε, κι όμως, ε, επειδή έχει θετικά αποτελέσματα στους ε, κατοίκους, ε, τελικά μπορεί να είναι α, αποδοτικό. Ενώ κάτι άλλο το οποίο δεν έχει καθόλου παρατυπίες, καθόλου λάθη, δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό. Παρότι δεν έχει λάθη. Επομένως, ας το αντιμετωπίσουμε, ας το αντιμετωπίσουμε αυτήν την μελέτη σαν ένα πρώτο βήμα. Ε, μιλάμε όμως για την αποδοτικότητα. Εδώ ε, έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές μεθόδους ε, μακροοικονομικές κτλ. Μιλάμε λοιπόν για παρατυπίες, λάθη και απάτες εν κατακλείδη. Να μας παρουσιάσετε και την τελευταία σας μελέτη. Την μελέτη για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην, ε, κάτω, στις κάτω χώρες, στο Ηνωμένο και στην Πορτογαλία. Okay. Non okay. Βεβαίως, τα έχετε πει. Ναι, έχουμε τελειώσει λοιπόν, αφού τελειώσαμε και με αυτό το σημείο. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Noi facciamo la riunione dei coordinatori adesso e con il resto della Commissione domani alle 9. Κοιτάξτε, α μείνουν μόνο οι συντονιστέ για τι συνεδρίες των συντονιστών τώρα και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού μπορούν να φύγουν. Θα τα ξαναπούμε στην πλήρη σύνθεση αύριο το πρωί στις 9.